Άρχεται λοιπόν η συνεδρίασή μας όπου θα έχουμε την παρουσίαση του κυρίου Μάριο Μόντι. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Θα μας παρουσιάσει μαζί με τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ομάδα υψηλού επίπεδου, τον Αλέλα Μασού, τον Κίφερ Χόφστατ, και τον Ιβάιλο Κάλφιν. Θέλω να χαιρετήσω που συμμετείχαν σε αυτές τις εργασίες της ομάδας εργασίας για τους ίδιους πόρους για τον προπολογισμό της Ένωσης. Για την ημερήσια διάταξη τα σημεία 4, 5 και 6 αναβάλλονται. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο από την πλευρά του Συμβουλίου. Πρόκειται για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 14-20. Η Ιταλία διατήρησε την επιφύλαξή της κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 13ης 12ου, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τα μέτρα που θα ληφθούν υπευθύνη της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας. Οι συντονιστές, κατά τη συνεδρίαση στις 8 Δεκεμβρίου, αποφάσισαν να ζητάξουν μια γνωμοδότηση για την έκθεση ΕΚΟΝ κοινή βάση για τον ε, ε, εταιρικό φόρο, για τον κοινό εταιρικό φόρο. Θα την αναλάβει η Σοσιαλιστική Ομάδα και στη συνεδρίαση της 9 Ιανουαρίου η ευρεία πλειοψηφία των συντονιστών εξέφρασαν την ε, άποψη ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ έχει τις αναγκαίες ε, ικανότητες για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτά ήθελα να σας πω σε ενημέρωση. Και τώρα να ακούσουμε τον Μάριο Μόντι. Υπογραμμίζω την πολιτική σημασία κεφαλαιόδη που είχε αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου το κοινοβούλιο μας και ιδιαίτερα η Επιτροπή Προϋπολογισμών οπωσδήποτε θα εργαστούν για να εφαρμόσουν τις προτάσεις της έκθεσης αυτής. Το πολιετές δημοσιονομικό 1420 έγινε δεκτό υπό μια διπλή επιφύλαξη να υπάρξει μια ενδιάμεση στη μέση της διάρκειας αναθεώρηση και η δεύτερη προϋπόθεση ήταν να μελετήσουμε ενδεχόμενους ίδιους πόρους για να αυξήσουμε την χρηματοδότηση του προπολογισμού. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Η τελική έκθεση της ομάδας ε, σας έχει σταλεί, αλλά δεν θα πρέπει να γνωστοποιηθεί πριν την ερχόμενη Τρίτη. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα γίνει γνωστό το περιεχόμενο εφόσον ε, είναι δημόσια αυτή η συνεδρίαση και ο Μάριο Μόντι θα παρουσιάσει στον τύπο την έκθεσή του αμέσως μετά την συνεδρίασή μας. Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν στις 11.30. Ο κύριος Φερχόφστατ και ο κύριος Μουρεσάν πρέπει να φύγουν στις 10 γιατί θα λάβει χώρα η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών για το θέμα των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Ευχαριστώ τον Ζίγφριντ Μουρεσάν που ε, θα με εκπροσωπήσει σε αυτή τη συνεδρίαση. Οπότε να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μάριο Μόντι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και για την εισαγωγή που κάνατε στην Επιτροπή ε, που προεδρεύετε έχετε ένα σημαντικό ρόλο και θα εξακολουθήσετε να έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως και η Επιτροπή σας ε, εμπνέοντας ε, και παρακολουθώντας την εξέλιξη των εργασιών. δεν συνάδει με τον αρχικό προγραμματισμό, αλλά σκόπιμο θα ήταν να πω ότι η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η έκτακτη αυτή συνεδρίαση, όπως λέει η μερίσια διάταξη, αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία για δημόσια συζήτηση αυτής της ε, έκθεσης και των συστάσεων της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους. Εξάλλου, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Προεπολογισμών καθορίζεται και αναγνωρίζεται διαρκώς και τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των ιδιών πόρων. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η χρηματοδοτική πλευρά του προπολογισμού πέραν τη πλευρά των δαπανών για την οικονομική αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πέραν αυτού γνωρίζετε επίση πολύ καλά πώ ε, αυτό επηρεάζει το, η θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την εμπιστοσύνη και την ε, νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά τις ικανότητες της να επιτύχει τους στόχους της και να υλοποιήσει τις πολιτικές της δεν είναι η σύμπτωση που η δημιουργία της ομάδας υψηλού επίπεδου ξεκίνησε από εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αξίζεται συγχαρητήρια μάλιστα, διότι εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίσατε ως μέλη της ομάδας αυτής Ορισμένες από τις εξέχουσες προσωπικότητες σας από όλους τους ε, τομείς ε, αλλά και ειδικευμένου σε αυτά τα ζητήματα και θα ήθελα να εκφράσω από βάθος καρδιάς την εκτίμησή μου προς τον Αλάν Λαμασούρ, τον Κίφερ Χοφστάτ και τον Ιβελο Κάλφιν Όλοι τους ε, συνέβάλαν ε, ενεργά, με υπομονή, με ενθουσιασμό στις προσπάθειες της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ε, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα και εσείς διαδραματίσατε ρόλο κλειδί σε πολλές δημόσιες συζητήσεις, σε πολλές διασκέψεις και ανέκαθεν δίνατε ένα μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, εκφράζοντα το εξαιρετικό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι δίθεσε στην ομάδα μα κάποιε διοικητικέ δυνατότητε και αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία ε, στην διοργανική γραμματεία υπήρξε πολύ επικοδομητική και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ρεαλιστές ε, και χάρη στην καλή θέληση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω κυρίως ε, τον επικεφαλής Αν ε, Μοντανιό της Task Force για τους ίδιους πόρους. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Η σύνθεση της ομάδας ε, χαρακτηρίζεται από προσωπικότητα σε ψηλό με διαφορετική εμπειρία ο καθένας, αλλά ουσιαστικά ο καθένας τους ε, έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πολιτικές ευθύνες ε, στα ευρωπαϊκά όργανα, στα κράτη-μέλη. και το γεγονό ότι το καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα διόρισε τρία μέλη στην ομάδα ε, σημαίνει ότι και οι ιδιαιτερότητε και οι ευαισθησίε του κάθε θεσμικού οργάνου έπαιξαν κάποιο ρόλο. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η αρμονία που δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ομάδας ε, ήταν εκείνη που οδήγησε, βοήθησε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα ουσιαστικά ομόφωνα. Καταλήξαμε σε εννέα συστάσεις, οι οποίες ε, έχουν εγκριθεί ομόφωνα, πέραν, με εξαίρεση μια μικρή υποσημείωση που θα βρείτε με μια διαφωνία ενό μέλους για μία από τις εννέα συστάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να το εισακούσουν τα τρία θεσμικά όργανα στις συζητήσεις τους, διότι μετά από τις ε, εντατικές ανταλλαγές απόψεων που χρειάστηκαν δύο χρόνια ε, και με πολλές εξωτερικές διαβουλεύσεις, φυσικά ο καθένας έδρασε βάσει των δικών του ιδιωτήτων, αλλά και υπεύθυνα ενώπιον ε, των θεσμικών οργάνων. Και έτσι καταλήξαμε σε ομόφωνες συμφωνίες ε, σε θέματα τα οποία παραδοσιακά είναι ιδιαίτερα επίμαχα, ε, ειδικότερα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Να στραφώ στα βασικά καταληκτικά μηνύματα της έκθεσης. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όχι επικρίνοντας ε, ότι δεν πήγαινε καλά με τους ιδίους πόρους, αλλά με τις καλές τους πλευρές, με τα πράγματα που λειτουργούν σωστά. Η εκθέσή μας περιλαμβάνει πολλές ε, συστάσεις, πολλά κεφάλαια για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικά διότι αποτυπώνουν την διοργανική μας συνένεση, τη διοργανική μας συμφωνία. Αν είχαμε επικεντρωθεί μόνο στις ελλείψεις, θα είχαμε έρθει σε σύγκρουση με πολλούς ε, ενδιαφερομένους ε, και θα είχαμε αποδυναμώσει τη δυνατότητα να μας πάρουν στα σοβαρά και να επιτύχουμε τελικά. Αντιθέτως, ε, υπογραμμίσαμε τα σημαντικότερα προνόμια του σημερινού συστήματος, στην αρχή της ισορροπίας που απαιτεί τον ισοσκελισμό πάντα του προϋπολογισμού, ε, το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που αποτέλεσαν το πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, τα ε, στελωνιακούς δασμούς ε, που αποτελούν υπόδειγμα για το τι πρέπει να είναι οι παραδοσιακή πόροι το πόρο που βασίζεται στο ΕΠ και τους υπολοιμματικούς ιδίους πόρους που αποτελούν ένα ευέλικτο και σταθερό ε, εισόδημα. οποιοδήποτε νέο πόρος που θα βασίζεται σε φόρο και που μπορεί να αντικαταστήσει, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις σημερινές συμβολές από το ΑΕΠ ε, έστω εν μέρη. Η προσέγγιση μας ήταν να διευρύνουμε την προοπτική πέραν ε, των ταμείων των κρατών μελών της υιοθέτησης προπολογισμών στις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο. Επίσης, θέλησαμε να διευκρινίσουμε ε, για το τι θα χρησιμοποιούνται οι διπόροι πέραν της απλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνοντας ε, τα πολιτικά ωφέλη. Ε, στην έκθεση υπάρχουν ενοιολογικές διευκρινήσει. Και εκεί δεν έχουμε μείνει ακαδημαϊκοί, σας διαβεβαιώ. Δεν έχουμε παραμείνει σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτές οι διευκρινήσεις μας βοηθούν να συνεχίσουμε το διάλογο για να ξεκινήσουμε αρχικά. Ε, πρέπει να πούμε ότι οι δίποροι δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, οι καθυστερημένες πληρωμές, ε, το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορούν να επιληθούν ε, αλλάζοντας απλά τους ε, τρόπους με τους οποίους αποκομίζουμε έσοδα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την ορολογία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Η έκθεση παρέχει ορισμένους ορισμούς εργασίας, περί του τι είναι ένας γενικός πορός εισοδήματος και ξεκαθαρίζει το νομικό καθεστώς των ιδιών πόρων. Η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας δεν είναι κάτι νέο. Δεν μπορούμε να την απορρίπτουμε ως κατευθυντήρια γραμμή διότι διότι έχει να κάνει με την νομιμότητα της ευρωπαϊκής δράσης. Ε, ξέρετε, το πιο πράγμα που είχαμε σε όλο αυτό το εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε, ήταν ότι μας ζητήθηκε να ερευνήσουμε την πλευρά των εσόδων ε, στο, πλαίσιο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και τις πολιτικές ε, εγγενείς σχέσεις μεταξύ αυτού του τμήματος και των υπόλοιπων εσόδων αλλά και μεταξύ της πλευράς των εσόδων και της πλευράς των δαπανών. Και σε τελική ανάλυση οι δεσμοί μεταξύ του προπολογισμού και του λόγου ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν αναπόφευκτα, αναδείχθηκαν αναπόφευκτα με μεγάλη σαφήνεια. Δεν προσπαθήσαμε να διευρύνουμε τη δική μας εντολή. Δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά είχαμε διακρίνει μια έκκληση και από τα τρία θεσμικά όργανα κάθε φορά που συναντιόμασταν για διαβουλεύσει ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή. Διότι δεν πρόκειται για άμεσα μόνο για το θέμα των ιδιών πόρων, αλλά διότι όλα συσχετίζονται μεταξύ του και παίζουν σημαντικό ρόλο στην συνολική εικόνα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η έννοια της ε, σωστής απόδοσης του Ζουστρετούρ θα πρέπει να ε, μείνει πίσω, να το αφήσουμε πίσω, να το ξεπεράσουμε, όπως και να ε, ξεφύγουμε από το διέξοδο που χαρακτηρίζει εδώ και καιρό όλες τις ζητήσεις περί προϋπολογισμού. Παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι όλοι κατανοούν από κοινού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τις πρόσφατες ε, σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ε, κινητοποίηση επενδύσεων ε, για θέματα όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση. Συμφωνούν όλοι ότι οι δαπάνες Ευρωπαϊκής πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά κοινοφιλή αγαθά. Αυτό θα μας οδηγήσει και στο μέλλον για, μια πιο κλασική, για ένα πιο κλασικό όραμα δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε μέχρι στιγμής δεν υπήρξε δεν θεωρήθηκε όργανο αναδιανομής αλλά θα μπορούσε θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μηχανισμό που θα παρέχει στους πολίτες μας αγαθά και υπηρεσίες δημόσιας φύσης πρώτον και δεύτερον δημόσιας φύσης που αδυνατούν να παρέχουν σήμερα τα κράτη-μέλη. Ό,τι είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικότερα όσον αφορά τι διάφορε κρίσει, η καθεμία από τι οποίε αντιμετωπίστηκε ω επίγουσα, αλλά οι οποίε ε, ταυτόχρονα αποτέλεσαν δομική επίγουσα, ε, δομικές επίγουσες καταστάσεις που μας ανάγκασαν να επανεστιάσουμε τον τρόπο σκέψης μας ε, ε, γύρω από τα δημόσια αγαθά που μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς, ε, ποιες είναι οι οικονομικές απαιτήσει ε, για κάτι τέτοιο. Οπότε αυτός ο ορισμός του δημοσίου, του αγαθού θα πρέπει να εξεταστεί πιο διεξοδικά στο άμεσο μέλλον και ένα από αυτά τα αγαθά θα είναι η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόσφατο άρθρο στον τύπο χαρακτήρισε την προσπάθειά μας, μια προσπάθεια να γίνουν λιγότερο τοξικές οι διαπραγματεύσεις του προπολογισμού μια αντίδραση στο δηλητήριο της επιστροφής της λεγόμενης, αλλά πρέπει βεβαίως να δούμε και το κοινό συμφέρον και τα ωφέλη που έχουμε, τα ωφέλη που έχουμε αντί να εστιάζουμε συνεχώς σε ροές και να ελαχιστοποιούμε τις εθνικές συνεισφορές αντί να επενδύουμε στο κοινό καλό. Και χάρηκα που άκουσα τον Επίτροπο Έτιγκερ να δίνει παραδείγματα νομίζω στην ακρόαση της προάλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κρατηδίου του της Βάδης Βίρτεμβέργης για το πώς επίσης ωφελείται άμεσα και έμεσα από την εσωτερική αγορά και την πολιτική συνοχής και τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης ε, των διαρθρωτικών ταμείων και σε άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή το σκεπτικό ότι οι έξυπνες επενδύσεις θα αποδώσουν αργά ή γρήγορα και ότι δεν είναι απλά ζήτημα αλτρουισμού, είναι κάτι το σημαντικό. Αλλά βεβαίως τα προγράμματα δαπανών πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Για να είμαι σύντομος ε, και με την άδειά σας ε, κύριε Πρόεδρε ε, επειδή θέλουν και οι τρεις συνάδελφοι στην ομάδα να συμπληρώσουν κάποια πράγματα δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για τους πιθανούς νέους ίδιους πόρους. Να πω μόνο ότι τους ε, ομαδοποιούμε, κάνουμε μια τεχνική ανάλυση του κάθε πιθανού νέου ίδιου πόρου και έχουμε πρώτον αυτοί που σχετίζονται με την ε, εσωτερική αγορά και τον φορολογικό συντονισμό και δεύτερον πιθανοί ίδιοι πόροι που σχετίζονται με την ενεργειακή ένωση, το περιβάλλον, το κλίμα και τα Θα τα αναπτύξουν ίσως οι συναδελφοί και το συμπέρασμα που θα ήθελα να σας αναφέρω αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρωί πριν από την συνεδρίαση έδωσα ένα αντίγραφο της τελικής έκθεσης και των συστάσεων στον πρόεδρο Σούλτς και συμφωνήσαμε ότι η δημοσίευση της έκθεσης Προφανώς δεν είναι το τέλος της ε, διαδικασίας, αλλά μπορεί να είναι το τέλος της δικής μας συνεισφοράς βεβαίως. Αλλά ελπίζω να αποτελέσει ένα ορόσημο και έναν καταλήτη στις ε, διαβουλεύσεις και θα ήθελα να επενέσω τα τρία θεσμικά όργανα γιατί ίσως ε, επί τη ευκαιρία εφήβραν μια νέα μορφή Συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων. Από όσο γνωρίζω ε, υπήρχαν πολύ γνωστές εκθέσεις που προετοίμασαν την νομισματική ένωση, την ε, αλλαγή των δημοσιονομικών κανονισμών ε, και των χρηματοπιστωτικών κανονισμών μετά την κρίση, αλλά από όσο γνωρίζω για πρώτη φορά έχουμε μια ομάδα η οποία είναι ταυτόχρονα πολιτική και τεχνική που συναισθήθη από κοινό από τα τρία όργανα και νομίζω πως ε, μπορεί χωρίς ε, να έχει την πολιτική ευθύνη κανένα από τα τρία θεσμικά όργανα να αποβεί ένα μοντέλο για να υπάρξει μια ελάχιστη συνένεση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, για την ε, συνεχή σας ε, στήριξη στις ε, προσπάθειές μας και ευχαριστώ την Επιτροπή Προϋπολογισμού για τον ρόλο που συνεχίζει να παίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας κατανοούμε όλη τη σημασία αυτής της έκθεσης και των προτάσεών της και στην ουσία περνάει τώρα η σκητάλη από την ομάδα αυτή στα τρία θεσμικά όργανα και αναμφίβολα το Κοινοβούλιο θα αξιοποιήσει αυτή την έκθεση για να προωθηθεί το θέμα αυτό, το ώστε ο προπολογισμό της Ένεσης να είναι ευανάγνωστος και κατανοητός όχι μόνο για τις κυβερνήσεις αλλά και για τους ε, πολίτες της Ένωσης. Προτείνατε οι τρεις συνάδελφοι που ε, ήταν επίσης μέλη της ε, ομάδας σας να πάρουν το λόγο. Να πάρει πρώτα, θα πρότεινα ο κύριος Γκί Φερχόφσταντ, γιατί πρέπει να φύγει για τη διάσκεψη των Προέδρων. Ο κύριος Φερχόφσταντ. Με συγχωρείτε που παίρνω το λόγο πριν από τους άλλους δύο συναδέλφους, τον Αλέν και τον ε, Άιβαλο. και να ξεκινήσω ευχαριστώ τον Μάριο Μόντι και νομίζω ότι εκφράζω την άποψη ε, ολόκληρης της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι Μάριο, εάν δεν προέδρευες εσύ, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα είχαμε μια τέτοια εκθέση, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη δυσχέρεια εκπόνησης μιας ε, τόσο αναλυτικής έκθεσης ε, για ένα τόσο λεπτό θέμα με συμμετοχή των τριών θεσμικών οργάνων. Η διαδικασία, όπως είπε και ο Μάριο, θα μπορούσε να είναι υπόδειγμα για άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ένωση δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει άλλη κατανόηση των απόψεων και αντί να έχουμε αντιπαράθεση από την πρώτη στιγμή να γίνεται προσπάθεια για να δούμε τι μας ενώνει. Δεύτερον, από πλευράς του Κοινοβουλίου, η έκθεση αυτή είναι βεβαίως ε, μια αφετηρία για το νέο πολιετές πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Αλλά πρέπει επίσης να θεωρηθεί και ως αφετηρία για τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit. Στο ψήφισμα που εκπονούμε αυτή τη στιγμή ε, για τις διαπραγματεύσεις αυτές για το Brexit που θα συζητηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και ίσως και το Μάρτιο και θα κριθεί βέβαια μετά την πυροδότηση του άρθρου 50 ένα τμήμα λοιπόν αυτού του ψηφίσματος θα ασχοληθεί ή θα βασιστεί στην έκθεση αυτή. Γιατί στην έκθεση έχουμε συμπεριλάβει και τις επιπτώσεις του Brexit. Και μία από αυτές είναι ότι δεν θα υπάρχει πλέον ε, Βρετανική επιστροφή. Οπότε δεν θα υπάρχουν και επιστροφές επί των επιστροφών. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική ε, δεν ισχύει πάντα η λογική. Αλλά αυτό καθιστά και την έκθεση αυτή τόσο ενδιαφέρουσα. Προτείνει μια ε, προσέγγιση για τον Brexit και για τις επιπτώσεις που θα έχει στο, στο επόμενο πολίτες πλαίσιο, για τις επιστροφές, τις επιστροφές επί των επιστροφών και για τα έσοδα. Επίσης, Πρέπει να περιορίσουμε επίσης και συμφωνώ ε, όλη αυτή τη συζήτηση για το juste retour όπως είπε και ο Μάριο. Γιατί. Ιδιαίτερα η σύσταση 4 λέει ότι ο πόρος που βασίζεται στο ΑΕΠ που στην ουσία είναι επιδότηση των κρατών προς την Ένωση δεν πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να περιοριστεί και πρέπει να αντικατασταθεί όχι από μία μόνο, από έναν μόνο ίδιο πόρο, αλλά από ένα σύνολο που να λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση, την παραγωγή και τη μόλυνση. Και αυτός, αυτή η δέσμη νέων ίδιων πόρων πρέπει να δημιουργηθεί, ούτω ώστε να δημιουργεί αυτομάτως μια ισορροπία στην πλευρά των εσόδων των κρατών μελών. Αν ε, λοιπόν λάβουμε υπόψη την παραγωγή, τότε κάποιες χώρες θα πρέπει να δίνουν περισσότερο στον προπολογισμό. Αλλά αν λάβουμε υπόψη την κατανάλωση, άλλες χώρες θα συμβάλλουν περισσότερο στον προπολογισμό της Ένωσης. Και αν λάβεις υπόψη την ε, μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε και πάλι μπορεί αυτό να επιβαρύνει άλλα κράτη-μέλη, δημιουργώντας λοιπόν μια δέσμη Συνδυάζοντας λοιπόν ε, τους ίδιους πόρους με αυτούς τους τρεις παράγοντες, παραγωγή, κατανάλωση, μόλυνση, δημιουργείς μια εξισορρόπηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία επιπλέον εξισορρόπηση. Είναι πολύ περιορισμένη. Και αν υπάρξει ένα σύστημα επανεξισορρόπησης, όταν χρησιμοποιείς αυτούς τους ίδιους πόρους, τότε πρέπει αυτό το σύστημα να είναι χρονικά περιορισμένο να καταργείται δηλαδή μετά από κάποιο διάστημα. Και γι' αυτό ε, θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που συχνά συμβαίνει στην πολιτική, ότι κάτι προσωρινό γίνεται μόνιμο. Και κάτι ακόμη. Βλέπω τον Αλένα να κοιτάζει τώρα το παράρτημα 4 της έκθεσης, οπότε μάλλον θα ασχοληθεί και εκείνος με αυτό το θέμα που θα αναφέρω τώρα. Στην έκθεση συμπεριλάβαμε και κάποια καθήκοντα, ότι πρέπει να επανέλθουμε στην ενότητα του προϋπολογισμού. είναι το παράρτημα 4, που είναι ένας πίνακας του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Γι' αυτό επιμείναμε να συμπεριληφθεί. Ορισμένα μέλη της ομάδας μας δεν ήθελαν να συμπεριληφθεί ο κύριος Μόν. Ναι, ναι, μα η αυτή στην έκθεση, η σελίδα αυτή στην έκθεση, οπωσδήποτε. Θα συμπεριληφθεί και στο αντίγραφο της έκθεσης που θα σταλεί στα άλλα όργανα. Συνεχίζει ο κύριος Φερχόστατ, βεβαίως ευχαριστώ τον Μάριο. Ήταν ε, μεγάλη τιμή που μπόρεσα για το θέμα αυτό να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντι που καθοδήγησε τις εργασίες αυτές. Από πλευρά μου, από μου δεν ήταν δύσκολο γιατί το περιβάλλον ήταν πολύ θετικό στην ομάδα. Όλοι εργαστήκαμε με το ίδιο πνεύμα, να βελτιώσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, να τον κάνουμε πιο υπόλογο, πιο διαφανή, πιο αποτελεσματικό. Και πιστεύω ότι αυτό οδήγησε στην ε, συμφωνία ε, που οφείλεται φυσικά και στην, ε, στον ικανότατο πρόεδρο και έτσι καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ήθελα καταρχάς επίσης να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο και στη Γραμματεία διότι ε, αυτά τα δυόμιση χρόνια πολλές φορές χρειάστηκε να γράψουμε εκθέσεις, να συντονίσουμε θέσεις ε, και εγώ ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στην ομάδα υψηλού επίπεδου ε, πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν πολύ χρήσιμο γιατί η ομάδα μας ενημερωνόταν τακτικά και γνώριζε τι συνέβαινε, πώς συνέβαινε κάτι το οποίο πάντα αποτελεί προϋπόθεση για ένα καλό αποτέλεσμα. Κάποια πράγματα ήθελα να πω, όχι τόσο για το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά ως τροφή προσκέψη. Ας θεωρήσουμε ότι το, η εκθέση αυτή είναι ένα σενάριο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ώστε να γίνει πιο διαφανής, πιο υπόλογος, ε, να την χάρει καλύτερη διαχείριση. Θέτει ως στόχο το 50% τουλάχιστον των ίδιων πόρων να προκύπτουν από επιπλέον πόρους και έχουμε διάφορες ε, προτάσεις για αυτούς τους επιπλέον πόρους με πολύ καλές ε, τεχνικές αναλύσεις της κάθε πρότασης. Αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτήν την έκθεση, όπως θα δείτε, ήταν να φτιάξουμε ένα σενάριο εφικτό, χωρίς αλλαγή της συνθήκης, χωρίς ε, μεταβολή εξουσιών, χωρίς ε, παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Ε, όλες οι ανησυχίες δηλαδή που συνήθως εκφράζονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια στα κράτη-μέλη έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την έκθεση. Οπότε όλα αυτά δεν αποτελούν πλέον ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι αυτό το σενάριο που προτείνουμε εμείς είναι εφικτό και ρεαλιστικό. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε στο μέλλον, αυτό εδώ είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αυτή η έκθεση, αλλά από μια έκθεση μέχρι να φτάσει κανείς στις πολιτικές υπάρχει πολλής δρόμος και το δρόμο αυτό θα πρέπει να διανύσουμε φυσικά συνεργαζόμενοι μεταξύ των ε, ε, οργάνων της Ένωσης, αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους εμπειρογνώμονες, ώστε αυτός ο πολύ σκοτεινός τομέας ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να γίνει πιο ξεκάθαρος ε, για τον κόσμο, να γνωρίζουν οι πολίτες τι πληρώνουν και τι λαμβάνουν για τους φορούς που πληρώνουν. Οπότε αυτή η συζήτηση για να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο και οι σχετικές πολιτικές θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές και τα Εθνικά Κοινοβούλια της Περιφέρειας και τους ε, όσους Τη υπευθύνους χάραξης απόψεων. Αυτό είναι το σενάριο λοιπόν, αλλά σκεφτούμε λίγο και πέραν αυτού. Αρκούν αυτά για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ θα έλεγα όχι. Αν δούμε ολόκληρο το σύστημα των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, συμπεριλαμβάνουμε των εθνικών προπολογισμών, του ευρωπαϊκού προπολογισμού και του ζητήματο που αναπόφευκτα θα προκύψει στι συζητήσει ε, τη δημοσιονομική ικανότητα τη ευρωζώνη σε σχέση με τον προπολογισμό. Στο τέλο, ε, οι φορολογούμενοι είναι οι ίδιοι, ξέρετε, οπότε καλό θα ήταν να διευρύνουμε λίγο τον τρόπο σκέψη μα και να δούμε πώ τα δημόσια οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καταβάλλονται από του ίδιου φορολογουμένους θα μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναπτύξουμε άλλο ένα σενάριο, το οποίο να μην αφορά μόνο του πόρου και τη βελτίωση του τρέχοντο προπολογισμού, αλλά να σκεφτούμε πέραν αυτού. Να σκεφτούμε πώς δεν θα επιβαρύνουμε περισσότερο τους πολίτες, πώς μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά οικονομικά, κάθε ευρώ που δαπανάται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή του εθνικού προπολογισμού να πηγαίνει στο σωστό σκοπό και να παρέχουμε στους πολίτες αυτό που αναμένουν. Τι μπορούμε να κάνουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχουμε κάποιες πολιτικές προστιθέμενες αξίες όπως η μεταναστευτική πολιτική ή την πολιτική ασφαλείας. η συντονισμένη προσπάθεια φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από ότι θα έφερνε προσπάθεια ενό επιμέρου κράτου μέλου, οποιοδήποτε κράτου μέλου. Οπότε πρέπει να δούμε, ξεκινώντα από το μηδέν, ε, πρέπει να δούμε τι εικόνα θα πρέπει να έχουν τα ευρωπαϊκά οικονομικά και εκεί δίθεται το σύνθεση ερώτημα. Οι εθνικοί ε, προπολογισμοί και ο συντονισμό του με τον ευρωπαϊκό, πώ αλληλοσυμπληρώνονται, τι ευελιξία απαιτείται και πώ κινητοποιείται ο ευρωπαϊκό προπολογισμό για την επίλυση προβλημάτων που αναδύονται ε, ειδικότερα αυτά που θα έχουμε μετά την υιοθέτηση αυτού εδώ. Εγώ θα ήθελα ένα πιο φιλόδοξο σενάριο, ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο ίσως απαιτεί κάποιες αλλαγές ε, στην συνθήκη και περισσότερες ε, πολιτικές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Δηλαδή, βασιζόμενοι σε αυτό, κάτι το οποίο είναι εφικτό, αυτό το οποίο προτείνουμε, Νομίζω πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω στην ανάπτυξη του ζητήματος των ιδίων όρων. Τέλος, κάτι για τον χρόνο. Ο Γκί μόλις ανέφερε το Brexit. Νομίζω πως έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αλλάξει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Και το θέμα του Brexit δεν είναι ε, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα είναι ήδη αρκετά δύσκολο από την ε, σκοπιά του προπολογισμού, αλλά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει λοιπόν να ε, απαντήσουμε στις ανησυχίες των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Βρετανοί ψήφισαν λάθος και έκαναν λάθος και παραπλανήθηκαν. Αν λοιπόν δεν γίνουν πιο κατανοητά τα δημόσια οικονομικά και ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός, κατά το οποίο σημαίνει τεράστιες μεταρρυθμίσεις, θα έχουμε το κείμενο να ε, μεταδοθεί αυτό το συνέστημα και σε άλλα κράτη-μέλη. Οπότε το Brexit είναι μια φορμή να σκεφτούμε. Τώρα δεν μου αρέσει η λέξη να πουλήσουμε, το πώς θα προωθήσουμε τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ε, πολίτες. Το ένα λοιπόν είναι η Brexit και ο άλλος παράγον είναι η προετοιμασία του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Από όσο ξέρω, φέτος η Κομισιόν θα αρχίσει ήδη να προετοιμάζει το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε ήδη συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν ξέρω εάν ε, ε, θα τα εγκρίνει αυτά. Αυτή η θητεία του Κοινοβουλίου είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί ίσως χρειαστεί χρόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα δούμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν πως αυτό τώρα είναι το παράθυρο της ευκαιρίας, από τώρα μέχρι την έγκριση του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, τα επόμενα δύο χρόνια, για να σκεφτούμε αλλαγές πιο φιλόδοξες, ή όχι τόσο φιλόδοξες, εάν δεν το επιτρέπει η πολιτική κατάσταση. Ε... Μάλιστα, και σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη στην έκθεση αυτή και θεωρώ πως είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσουμε τα δημοσιοοικονομικά. Ευχαριστώ, Αλένα Μασούρ. Ευχαριστώ. Και εγώ ε, χαιρετίζω την εργασία του Μάριο Μόντι και δεν είναι θέμα τυπικής ευγένειας. Όλοι όσοι συμμετείχαμε στις εργασίες ξέρουμε ότι χωρίς εκείνον δεν θα καταλήγαμε σε αυτό το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε όπως ε, ήδη αναφέρθηκε ε, με ομοφωνία μόνο μία μικρή επιφύλαξη, μία υποσημείωση για μία πρόταση ενός μέλους. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα είναι ότι θα διαπιστώσετε στις συστάσεις που κίνονται περιλαμβάνονται οι προτάσεις που εδώ και χρόνια έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνονται πολλές προτάσεις και στο πνεύμα και στη διατύπωση των επισήμων προτάσεων που έκανε ο Γιάννους Λεβαντόφσκι ως Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013 και λοιπόν τώρα οι προτάσεις αυτές δεν δεσμεύουν μόνο το Κοινοβούλιο ή την Επιτροπή. Είναι αποτέλεσμα των εργασιών μιας ομάδας όπου εκπροσωπεί το και το, κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο. Συγγνώμη. Το Συμβούλιο το οποίο είχε αρνηθεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό το 2013, τώρα όμως είναι υποχρεωμένο να το συζητήσει, ιδιαίτερα στα πλαίσια των επομένων πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Το θέμα αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. Και δεν το έχουμε αναφέρει στις συζητήσεις που έχουμε κάνει για τα βασικά ευρωπαϊκά θέματα μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και περισσότερες, ε, περισσότερη διάθεση για να αναπτύξει πολιτικές και πολιτικές μάλιστα οι οποίες να έχουν παγκόσμια επίπτωση με πενταροδεκάρες. Και είναι πολλά χρόνια τώρα που το λέει το Κοινοβούλιο αυτό. Και χρειάστηκε πρώτα απ' όλα η Επιτροπή Προπολογισμών να πείσει το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα καταφέραμε να γίνει αυτή η συζήτηση και σε επίπεδο Συμβουλίου γνωρίζοντας ότι για θέματα φορολογικά και δημοσιονομικά το, το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει με ομοφωνία αν θα γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο, αλλά η γνωμοδότηση αυτή δεν δεσμεύει πολιτικά το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι τώρα αρχίζει η πολιτική αντιπαράθεση. Σε ένα κλίμα γενικό που σε όλες τις χώρες όπως υπενθύμησε ο Γκί και ο Ιβάιλο ένα κλίμα όπου υπάρχει διαδεδομένος ε, ευρωσκεπτικισμός, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν θα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, το θέμα είναι πολύ λεπτό. Εάν κάποιος πολιτικός στην ίδια φράση αναφέρει τις λέξεις Ευρώπη και προπολογισμό, δεν νομίζω ότι θα αρχίσουν να τον αγκαλιάζουν και να τον φυλάνε. Και νομίζω ότι η αυτόματη στάση όλων των πολιτικών αλλά και των μέσων της κοινή γνώμης συνοψίζεται στο εξή. Αν θέλετε να αυξήσετε τον προπολογισμό της Ένωσης θα ε, επιδεινώσετε τη φορολόγηση των πολιτών. Γιατί πάντα οι φορολογούμενοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε αύξηση του προπολογισμού. Οπότε, εγώ θέλω εδώ στην Επιτροπή μας να στείλω αυτό το μήνυμα ότι μέσω την, ε, των εργασιών της ε, ομάδας αυτής καταλάβαμε ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη πολιτική διάσταση. Δεν ήταν ε, βέβαια στα πλαίσια της εντολής μας, αλλά πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε μια πολιτική πρωτοβουλία. Πρέπει να καταδείξουμε ότι ένα παραπάνω ευρώ που δαπανάται στις Βρυξέλλες επιτρέπει την εξοικονόμηση ενός ευρώ και πάνω στις εθνικές πρωτεύουσες που δαπανάται από τους εθνικούς προπολισμούς. Αυτή είναι η δημοσιονομική έκφανση της αρχής της επικουρικότητας. Και αυτό είναι και ένα έλλειμμα των συνθήκών μας. Καθορίσαμε στις συνθήκες την αρχή της επικουρικότητας. Στη συνθήκες της Λισαβόνας ε, περιλαμβάνεται και μια διαδικασία που επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να εξακριβώσουν εάν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας με αυτή τη διαδικασία κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, αλλά εφαρμόζεται μόνο για θέματα νομοθετικά. Μέχρι στιγμής κανένα θεσμικό όργανο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε κατά περίεργο τρόπο η Επιτροπή του το Κοινοβουλίο μας δεν έχουν ασχοληθεί. Κανένα θεσμικό όργανο δεν έχει ασχοληθεί με τη δημοσιονομική διάσταση τη αρχή τη επικουρικότητα. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που να λέει ότι όταν αποφασίζουμε, για παράδειγμα, ότι από, από τούδε και στο εξή, θα έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευση. Όπω προβλέπουν οι συνθήκε. Και όπω εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε σε περίπλοκε και καμιά φορά χαόδη συνθήκε, όταν λοιπόν λαμβάνουμε μια τέτοιου τύπου απόφαση, πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίζουμε ότι δεν δίνουμε μόνο την αρμοδιότητα στην Ένωση, αλλά και τους πόρους. Τους πόρους και από πλευράς ε, πιστώσεων και από πλευράς προσωπικού για να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα. Γιατί αλλιώς μετά Υπάρχει απογοήτευση από την κοινή γνώμη. Α, λένε οι Άγγλοι, Don't, Europe does not deliver. Παίρνουμε αποφάσεις, ε, καθορίζουμε στόχους, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ε, οι πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, είτε δεν συμβαίνει τίποτα, είτε γίνονται πολύ λίγα και με μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε η πρόταση που κάνω είναι πρέπει πάντα να διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά που δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, ένα φορέα, μια υπηρεσία, όταν για παράδειγμα δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να την πρικοδοτούμε με τις αναγκαίες αρμοδιότητες πρώτα απ' όλα για να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της, αλλά επίσης πρέπει να διασφαλίζουμε ότι σε εθνικό επίπεδο και ενδεχομένω και υποεθνικό, περιφερειακό, μειώνονται αναλογικά οι πόροι. Μέχρι στιγμή δεν έχει συμβεί καθόλου κάτι τέτοιο. Όταν δημιουργήσαμε την υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ένωση, φροντίσαμε να έχει το αναγκαίο προσωπικό. Έγινε 3-4 άτομα, ιδιαίτερα διπλωματικοί, αλλά σε μια χώρα, μεγάλη χώρα τη Ένωση που γνωρίζω καλά, ο υπουργό Εξωτερικών εγγυήθηκε ε, στι Ενώσει των υπαλλήλων του ότι δεν θα χανόταν ούτε μία θέση εργασίας. ενώ δημιουργεί μία νέα ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία. Επικάλυψη. Πρόεδρος. Και εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών, όταν προσπαθούμε να αγοράσουμε κτίρια για την υπηρεσία εξωτερική δράση στο Πεκίνο ή στο Τόκιο, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε μια 29η πρεσβεία στο Τόκιο και στο Πεκίνο. Βεβαίω, λέει ο κ. Λαμασούρ, θέλουμε να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και ένα ενιαίο, ένα και μόνο δίκτυο ευρωπαϊκή διπλωματία, αλλά διατηρούνται και τα εθνικά δίκτυα. Άλλο παράδειγμα, μια μικρή χώρα, δεν θα την ονομάσω, που εθίγει πολύ από την οικονομική κρίση του 2008 και 2009 και γι' αυτό κατήργησε τέσσερι πρεσβείε τη και μόλι επανήλθε η οικονομική κατάσταση, τι επανέφερε. Που δεν παίζουν κανένα ρόλο Επίσης, ένας από τους κύριους στόχους όταν είχαμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ήταν, ήταν να υπάρξει συνένωση των προξενικών μας υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε αφρικανικές χώρες εάν για ιστορικούς λόγους μία χώρα είχε προξενική παράδοση κτλ αν είχε προνομιακές σχέσεις με αυτή τη χώρα ή οι πρόξενοι αυτής, αυτής της χώρας να ασκούν προξενικά καθήκοντα για τις 28 χώρες. Και αυτό ξεχάστηκε εντελώ. Η Frontex. Αυξήθηκε ο προπολογισμό της, πήγε σε 500 εκατομμύρια. Για να είναι μια ευρωπαϊκή φυλακή. Πρέπει λοιπόν σε αντιστάθμιση του προσωπικού που θα δοθεί σε, σε αυτήν τη Frontex να μειωθούν αντίστοιχα οι εθνικές συνοριοφυλακές. Αλλά κανείς δεν το προτείνει αυτό. Και φυσικά οι εθνικές διοικήσεις θα επιδείξουν ιστερική εχθρότητα ε, μέσω των ενώσεων των υπαλλήλων. Οι υπουργοί επίσης ε, θα είναι αντίθετοι αλλά παράλληλα πρέπει να ε, φροντίσουν ε, οι δαπάνες τους να έχουν αποτέλεσμα και πολλοί τους άλλους υφίστανται πιέσεις για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά, άρα τους δίνουμε ένα καλό επιχείρημα. Τους λέμε ναι θα μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί κάποιες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στις Βρυξέλλες άρα αντικαθίστανται από ενωσιακούς υπαλλήλου. και οι καλύτεροι εθνικοί υπάλληλοι θα έχουν ε, την προοπτική απασχόληση σε ενωσιακό επίπεδο και όχι να παραμένουν σε εθνικό επίπεδο. Ήδη αναφέρθηκα ότι κάτι τέτοιο γίνεται για το άσυλο και τη μετανάστευση. Μέχρι στιγμής κανένα κράτος μέλος δεν επιχειρηματολογεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν τα κράτη-μέλη να αποδέχονται τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ένωση στα πλαίσια των συνδικών. Γιατί όλες οι προτάσεις μας ε, Ήδη υπόθηκε, σέβονται πλήρω τι συνθήκε. Είναι λοιπόν σαν τα κράτη-μέλη να δέχονται τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά να θέλουν να διατηρούν τους πόρους οικονομικούς και ε, ε, υπαλληλικού για να ασκούν αρμοδιότητες που δεν έχουν πλέον. Πρέπει να τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Αν θέλουμε να μα στηρίξει η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε στις Βρυξέλλες σημαίνει τουλάχιστον ένα ευρώ εξοικονόμηση από τους εθνικούς προπολογισμού. Και θεωρώ ότι, όπως ξέρει πολύ καλά η Επιτροπή μας και ιδιαίτερα ο κύριος Γκάιερ, μπορεί να είναι οικονομίες 28 ευρώ. Ένα σε κάθε χώρα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια διαδικασία. Δεν ξέρω, θα πρέπει να εμπλακούν και τα ελεκτικά συνέδρια των κρατών μελών, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ούτω ώστε να υπάρξει αυτή η δημοσιονομική διάσταση τη επικουρικότητας. Οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αυξάνουμε τους πόρους. Και με στόχο, αυτή πραγματικά είναι η φιλοσοφία τη επικουρικότητας, με στόχο ότι ορισμένε, όχι όλε, ορισμένε, όπω προβλέπονται από τι ηθίκες, βασιζόμεθα στι συνθήκε, εάν ασκούνται λοιπόν ορισμένε αρμοδιότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι ε, που θα ασκούνται πιο αποτελεσματικά από ό,τι αν ήσαν σε εθνικό επίπεδο. με Η αποστολή σας αφορούσε τους ιδίους πόρους. Ε? ώστε να θεραπεύσουμε την δημοσιονομική ε, αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά όταν μιλάμε για ιδίους πόρους πρέπει να μιλήσουμε και για δαπάνες φυσικά. Ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή σας, ε, τις παρουσιάσεις σας, ε, όλους τους προσκεκλημένους και να δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Και καταρχάς τους δύο μόνιμους εισηγητές μας για τους ιδίους πόρους, τον Γιάννος Λεβαντόφσκι, διευκρινίζοντας ότι λόγω απρόβλεπτων ε, ε, περιστάσεων δεν έχουμε μετάφραση από τα πολωνικά. Δεν θα διαμαρτυρηθώ. Κάπως θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις σας ε, και για την δύσκολη αποστολή που φέρατε εις πέρας από τις δυσκολότερες που μπορώ να φανταστώ ε, ειδικά δεδομένου του κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και βεβαίως σημασία έχει και η αξιολόγηση του τρέχοντος ε, συστήματος ε, το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά σε σχέση με τις ε, συνεισφορές με βάση το ΑΕΠ και βεβαίως πρέπει να δώσουμε προσοχή και στο ότι διαφέρουν τα λογιστικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε είναι δύσκολες οι συγκρίσεις μεταξύ κρατών. Αυτό το οποίο είναι χρήσιμο είναι αυτή η ευρύτερη έννοια της προστιθέμενης αξίας γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το καθεστώς της επιστροφής και τη συζήτηση ενό προπολογισμού των Βρυξελών. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε το πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν οι διάφορες πιθανές πηγές εσόδων γιατί εδώ πέρα βεβαίως έχουμε τη σύγκριση με την παρουσίαση που κάναμε το 2011 με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες υποθέσεις εργασίας, ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της συνθήκης ή αύξηση των ε, χρεώσεων των βαρών. Ε, εμείς οι παλαιοί με τον ε, Στέφαν Λένερτ βεβαίως τα είχαμε πει, φόρους στα καύσιμα, τον ηλεκτρισμό που αναφέρθηκε το 2011 και βεβαίως σε αυτά προσθέθηκε η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, τις νέες ε, εξελίξεις ε, για τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αφορούν την ασφάλεια, τη μετανάστευση, εξωτερικές ευθύνες, τα οικονομικά μέσα που βεβαίω υπάρχουν πλέον περισσότερα από το 2011, το ΕΦΣΙ, τα καταψεύματα και ο προπολογισμό του ευρώ. Το Brexit θεωρείται και μια ευκαιρία και έτσι το θεωρώ και εγώ, τουλάχιστον για απλοποίηση της πλευράς των εσόδων. Όμως, ε, βεβαίω χάνουμε ένα, μια εισφορά 5-6 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Αυτή ήταν η καθαρή εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπίζω μετά το 2020 οι συστάσεις είναι αρκετά προσεκτικές, ρεαλιστικές, αλλά ε, το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Έχει δίκιο ο Αλέν και ο Μάριο εδώ πέρα. Και η πολιτική βεβαίως αφορά και την εικόνα που υπάρχει. Και μόνο η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών δαπανών και η προστιθέμενη αξία του προπολογισμού θα βοηθήσουν να προχωρήσουμε στο να βρούμε νέες ε, πηγές εσόδων και να φύγουμε από τη συνεισφορά του με βάση το ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τι προσπάθειές σας και αποστολή εξετελέστη. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα έχει φτάσει η ώρα της πολιτικής. Σας ευχαριστώ, Ζαντεπρέ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι υπόλοιποι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντι και όλους τους συμμετέχοντες, διότι η ποιότητα του εγγραφού αυτού δεν σχετίζεται μόνο με την ευθεία του Προέδρου, αλλά και με τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό όλων των συμμετεχόντων. Ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, γιατί είναι σπάνιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο υψηλή ήταν η τεχνική ποιότητα του εγγράφου αυτού, ε, χωρίς ωστόσο να γίνεται δυσνόητο. Δεν χρειάζεται κανείς να γνωρίζει τέλεια την ευρωπαϊκή ορολογία για να καταλάβει ε, το ε, περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Οπότε σας ευχαριστούμε που συντάξετε ένα έγγραφο υψηλού τεχνικού επίπεδου και ταυτόχρονα πολύ ευανάγνωστο. Ήθελα επίσης ε, να χαιρετήσω την πολιτική ευφυΐα που χαρακτηρίζει αυτό το έγγραφο, το ρεαλισμό που το χαρακτηρίζει καθώς μένουμε εντός των συνθήκων και δεν μιλάμε αμέσως για τροποποίηση των συνθήκων με όλα τα προβλήματα που θα δημιουργούσε αυτό και όπως είπαν και οι προελίσσαντε, επιμένοντας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ουδετερότητας. Δηλαδή χωρίς καμία άμεση εφαρμογή ε, αύξησης ε, του φορολογικού άχθους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και επίσης Καλό είναι που υπενθυμίζουμε διαρκώς τι είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά πόροι. Είναι πόροι που κινητοποιούνται για την εφαρμογή πολιτικών και η συζήτηση που θα κάνουμε για τους ιδίους πόρους ε, δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ουσιώδη συζήτηση για τη φύση των ευρωπαϊκών πολιτικών και ειδικότερα των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών που πρόκειται να υλοποιηθούν. Τέταρτον, Πιστεύω ότι είναι, επίκαιρο φυσικά το έγγραφο, το είπαν όλοι, όχι μόνο γιατί θα οδηγήσει στη διαπραγμάτευση ε, μιας ε, ε, νέας κοινή δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και γιατί ε, θα θέσει ένα πρόβλημα το οποίο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Και τώρα, απευθυνόμενο στον πρόεδρο και στους συμμετέχοντες, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, το οποίο δεν εξετάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση, το ρυθμό υλοποίηση. Συμφωνούμε όλοι ότι η διαπραγμάτευση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Brexit θα πρέπει να επαναφέρει το θέμα ε, των ιδίων πόρων σε όλες τις συζητήσεις ε, που θα πρέπει να αποτελέσει ένα απόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε ζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά του ίδιου πόρου, ε, απευθύνω το ερώτημα μου στον κύριο Μόντι και στον κύριο Λεβαντόφσκι μπορούμε να φανταστούμε ότι θα είναι προοδευτική η εφαρμογή του μηχανισμού των ιδιών πόρων και να εξηγήσω ότι ενώ το Brexit θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων. Για να αντισταθμιστεί αυτή η μείωση των εσόδων μπορούμε να κινηθούμε είτε προς την αύξηση του συμβολής ε, των κρατών μελών από το ΑΕΠ ή με ένα σύστημα ιδιών πόρων. Επίσης, στο πίσω αυτού του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ότι οι νέες πολιτικές ε, και τα σχετικά κονδυλία να χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους. Δεν λέμε λοιπόν στα κράτη-μέλη ότι από τώρα α, διακόπτουμε τις ε, ε, συμμετοχές από το ΑΕΠ, απλά λέμε ότι θα βάλουμε μια νέα μηχανική που σιγά σιγά θα ενδυναμωθεί ε, όχι μόνο για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες από το Brexit αλλά και χρησιμοποιώντα ίδιου πόρου για τη χρηματοδότηση των νέων πολιτικών, για την αύξηση των ε, κονδυλίων ε, για υπάρχουσε πολιτικέ που θεωρούμε ότι είναι πολιτικέ υψηλή προτεραιότητα. Αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνω προ τον κύριο Μόντι και στα μέλη του πάνελ. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί προοδευτικά το σύστημα αυτό των ιδίων πόρων. Τέλος, ε, σε μία παραγραφή που διάβασα επιμένετε στο ότι από σήμερα ήδη πρέπει να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε όλους τους πόρους με τους οποίους δεν έχει ασχοληθεί ο φάκελος τους νέους ε, ε, ίδιους πόρους και πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ άριθμοι όχι μόνο αυτή που περιλαμβάνεται στο Η Κομισιόν τώρα προτείνει ένα σύστημα ε, προηγούμενης έγκρισης για όλους τους αλλοδαπούς ε, που θέλουν να εισέλθουν στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάθηκε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε ας πούμε αυτή η, προηγούμενη έγκριση θα κοστίζει 10-15 ευρώ οτιδήποτε. Η διαχείριση των κοινών συνόρων ε, γίνεται από τα κράτη-μέλη αλλά είναι κοινά τα σύνορα και τα έσοδα από εκεί μπορούν να τροφοδοτήσουν τον προπολογισμό της Ένωσης. Διότι πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε μια γενική αρχή ότι όλα τα άμεσα έσοδα που προέρχονται από την άμεση υλοποίηση των πολιτικών αρμοδιότητας τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας σχετικά απλός μηχανισμός και υλοποιήσιμος. Οπότε κύριε Πρόεδρε και μέλη του πάνελ, μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν κάποια δυναμική υλοποίηση, αλλά όχι υπερβολικά γρήγορη ενός πλήρου συστήματος και να προσανατολιστούμε επίσης στην αναζήτηση μιας γενικής αρχής που μπορεί να μας οδηγήσει να ανακαλύψουμε και άλλους πώς που δεν έχουμε φανταστεί μέχρι στιγμής ε, και να ενδυναμώσουμε αυτό το σύστημα των πόρων σιγά σιγά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα, περάσουμε, θα δώσουμε τώρα το λόγο στους συντονιστές των ομάδων. Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που πρέπει να τεθεί είναι πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την θαυμάσια εργασία της ομάδας αυτής που της οποίας προείδρευσε ο Μάριο Μόντι και την ε, ομοφωνία που επέτρεψε να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε τον προπολισμό της Ένωσης. Γιατί πάντα θέλουμε να σεβόμεθα τους ε, στόχους μας. Όμως ε, περιοριζόμεθα σε αυτό το περιορισμένο Μήμα του ΑΕΠ. Και έτσι απογοητεύουμε τους ε, πολίτες μας. Δίδεται η εντύπωση ότι με τους στόχους που έχουμε καθορίσει για το, την Ευρώπη 2020 θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, ε, των περιφερειακών ανισοτήτων. Όλα αυτά με 1% του ευρωπαϊκού ΑΝΕΠ. Εάν μείνουμε σε αυτήν την ε, ποσότητα σε αυτό το τμήμα, θα πρέπει καλύτερα να καθορίσουμε τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους περιορισμένους πόρους. Το θέμα των ιδίων πόρων. Θεωρώ ότι πρέπει να μπορεί να γίνει κατανοητό από την κοινή γνώμη για να μπορέσουμε να έχουμε την ευνοϊκή της αντιμετώπιση. Οπότε είναι θεμελιώδες το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Είναι δύσκολο όμω να καθορίσουμε. Εγώ τουλάχιστον ε, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να καταδεικνύουμε πάντα ότι ένα ευρώ του ευρωπαϊκού προπολογισμού σημαίνει κέρδος. Γιατί, γιατί το θετικό αποτέλεσμα ε, πολύ συχνά ε, έρχεται με μεγάλη διαφορά φάση. άρα δεν είναι εύκολο να φανεί ότι υπάρχει εξοικονόμηση, ότι μάλιστα ότι ένα ευρώ του ευρωπαϊκού προπολογισμού σημαίνει ότι έχουμε κέρδη ενός ευρώ σε κάθε εθνικό προϋπολογισμό. Ορισμένες φορές πρέπει να κάνουμε την ε, ε, απόδειξη με τον αντίστροφο πρώτο. Να πούμε δηλαδή ότι εάν δεν δαπανηθεί αυτό το ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει επιπτώσεις αρνητικές συνολικότερα για την Ένωση. Πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν τι σημαίνει ε, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Για παράδειγμα, πόσο κοστίζει η επίλυση της ε, προσφυγικής κρίσης, αλλά πόσο θα κόστιζε εάν δεν επιλύεται. Έτσι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει σύντομα. Αλλά σύντομα έχουμε εκλογές στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Και αυτό αποτελεί ακριβώς εμπόδιο στον ε, ουσιώδη διάλογο που θα έπρεπε να έχουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των ίδιων πόρων. Οι ίδιοι πόροι πρέπει, η συζήτηση για τους ίδιους πόρους πρέπει να συμβαδίζει με την προσπάθεια απλούστευσης του προπολογισμού, τόσο ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος. Ε, πρέπει να συνδυαστεί με το θέμα των επιστροφών. Είναι καλή ευκαιρία λοιπόν τώρα νομίζω να ε, απαλληφθούν όλες αυτές οι επιστροφές. να απαλληφθούν εντελώ. Κάτι άλλο. που έχει να κάνει και με αυτό που μόλις είπε τώρα ο συνάδελφος Ζεράν Ντουπρέμ. Κάτι που μπορούμε να αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο ακριβώς το e-εμπόριο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, το e-trade σημαίνει απώλεια πόρων για τα κράτη-μέλη. Αν όμως κάνουμε βήματα για να υπάρξει μια φορολόγηση του e-trade σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό να είναι ενωσιακός πόρος, θα μπορούσαμε να μειώσουμε την, ε, τα διαφυγόντα κέρδη. Αλλά θα έπρεπε φυσικά να υπάρξουν κάποιε επιστροφέ στου εθνικού προπολογισμού για την απώλεια παρόλα αυτά ε, πόρων ε, λόγω λιγότερων ε, εσόδων από τον ΦΠΑ. Είναι σαφές ότι αν δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε τις συνθήκες έχουμε μία πρόταση που σημαίνει πως δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να υποστούν επιπλέον φόρους. Αυτό πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή μας, η αποδοτικότητα των ενεργειών μας. Και πώς θα παρουσιάσουμε ακριβώς ε, τις προτάσεις αυτές για να επιτρέψουμε η συζήτηση για τους ίδιους πόρους να είναι συζήτηση για τις προτεραιότητες, για τις νέες πολιτικές και όχι να είναι συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει περισσότερα και πόσα θα επιστραφούν. Η συζήτηση για την πολιτική χρήση αυτών των ίδιων πόρων θα μας επέτρεπε να αποφύγουμε τη ζήτηση για το ποιος είναι καθαρός νησφορέας και ποιος ε, ε, ωφελείται από τον προπολογισμό. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση, καταδεικνύοντας ότι οι πολιτικές είναι αυτές οι οποίες βοηθούν συνολικά την Ένωση. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες που ε, ζητούν τέτοιες απαντήσεις. Εδώ και πολύ καιρό. Συγχαίρω λοιπόν ε, ε, τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτήν την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να δημιουργηθούν γνήσιοι ήδη πόροι στα πλαίσια της συζήτηση για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η κυρία Θάβαλ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντι που προείδρευσε των εργασιών αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου και όπως είπαν ήδη πολλοί, χωρίς τη δική του συμβολή, χωρίς τη δική του σωστή διεύθυνση των εργασιών, όπως ακριβώς μας είπαν ε, τα άλλα μέλη, δεν θα είχαν καταλήξει σε αυτά τα σωστά συμπεράσματα σε αυτό το κείμενο που περιέχει πολλή πληροφόρηση, πρέπει να την μελετήσουμε αναλυτικά όπως είπε και ο κύριος Μόντι η εντολή του ήταν να μελετήσει ένα τμήμα των ίδιων πόρων, αλλά τελικά αυτό το τμήμα των ίδιων πόρων έχει να κάνει συνολικά με τους πόρους της Ένωσης, έχει να κάνει και με τις δαπάνες, γι' αυτό η μελέτη τελικά διεύρυνε το, το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε και ευχαριστώ επίσης και τους τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάντα μας ενημέρωναν τακτικά όλα τα μέλη και τη Επιτροπή μα και του Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανταλλαγέ απόψεων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τη Επιτροπή, να ανταλλάσσουμε ιδέε, προτάσει, αμφιβολίε κτλ. Ούτω ώστε τελικά να έχουμε αυτό το τόσο αναμενόμενο κείμενο και θα αρχίσουμε να εργαζόμεθα επ' αυτού. Τώρα γι' αυτό το ζούστερο του, τη δίκαια επιστροφή. Σωστό είναι αυτό που υπόθηκε ότι θα πρέπει να βγάλουμε το δηλητήριο από αυτή την έννοια και τη ζήτηση για αυτή την έννοια. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη περισσότερο πρέπει να γίνει πιο σωστή συζήτηση. Αυτή η έννοια του juste retour είναι αυτό που δημιουργεί ε, πολλές ανησυχίες ε, στα πλαίσια της ε, προσπάθειας καθορισμού του πολιετούς πλαισίου, αλλά όταν συζητάμε τους ετήσιους προπολογισμού ούτε καν ασχολούμεθα με αυτό. Κάθε κράτος μέλος έρχεται με ένα χαρτάκι, ένα νούμερο που λέει εγώ δεν μπορώ να δώσω στον προπολογισμό πάνω από αυτό. Και δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικέ. Εγώ αυτό το ποσό έχω βάλει στον εθνικό προπολογισμό ω ε, μέγιστο που μπορώ να δώσω και θεωρούν ότι είναι δαπάνη, όχι επένδυση. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Από τη μία λοιπόν έχουμε το όριο του Ζήστρετουρ και από την άλλη έχουμε την προσπάθεια ελάχιστη συμβολή στου ενωσιακού πόρου και τον ενωσιακό προπολογισμό. Αυτό πρέπει να μα απασχολήσει σε όλη τη συζήτηση για του ε, ίδιου πόρου. Να αποφύγουμε αυτέ τι ε, πραγματικά στρεβλέ συζητήσει που δεν μα επιτρέπουν να έχουμε αρκετό χρόνο για να ασχοληθούμε με το τι ακριβώς πρέπει να περιέχει ο προπολογισμό πώς πρέπει να δαπανηθεί. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα του κ. Λαμασούρ για την επικουρικότητα. Και αυτό το τμήμα ότι πρέπει να λαμβάνει την υπόψη και στον προπολογισμό η επικουρικότητα. Και αυτό συνδέεται με τη δεύτερη μου ιδέα το ύψο του προπολογισμού. Αυτό ξέρω πω είναι ακόμη περισσότερο ταμπού από ότι του ίδιους πόρους. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Έχουμε τόσες προκλήσεις ενώπιόν μας, τόσες ανάγκες. Δεν επαρκεί το 1% του ΑΕΠ. Νομίζω ότι εφόσον συζητάμε για περισσότερους ίδιους πόρους, θα πρέπει να, κάνουμε, να μας επιτρέψει να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω σε αυτή τη συζήτηση. Οι δημόσιες επενδύσεις που χρειάζεται η Ένωση το προσφυγικό που έχει εκραγεί και δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Και για λόγους πολιτικής και για λόγους οικονομικούς. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προκλήση στην ενέργεια και την άμυνα που είναι μία από τις νέες μεγάλες προτεραιότητες της Ένωσης. Όλα αυτά δεν λύνονται με μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων. 1% του ΑΕΠ ούτε καν το 1,23 το οποίο μπορούμε να εγγύσουμε τώρα. Δεν επαρκούν όλα αυτά για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις ενώπιών μας. Και επιπλέον, φοβάμαι ότι κάποιες ε, πλευρές ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μόνο με την ε, πλευρά των δαπανών του προπολογισμού και να τροποποιήσουν κάποια κατανομή των, ε, των δαπανών για να αποφύγουν να ασχοληθούν με το άλλο τμήμα. Και η επιθυμία μου είναι να μην είναι και αυτή η έκθεση μία από τις θαυμάσιες εκθέσεις που εκπονούμε κάθε τόσο και μόλις δημοσιευθεί μετά την πετάμε στα αρχεία και δεν την ξαναβλέπουμε 30 χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να την έχουμε πάντα μπροστά μας και η Επιτροπή μας με βάση αυτήν να επιχειρήσει πραγματικά η Ένωση να καταλήξει στον προπολισμό που χρειάζεται και που θα αποδείκνει σε πολλούς ευρωσκεπτικιστές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θαυμάσια προσπάθεια της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα είναι και η προσθέμενη αξία τη Επιτροπή Προπολογισμών, ξέρετε. Ο κύριο Κόλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντι και την ομάδα εργασίας για την έκθεση αυτή. Και νομίζω πως η έκθεση αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας ε, να συζητήσουμε ουσιαστικά για όλα τα θέματα του προϋπολογισμού. Να συζητήσουμε σημαίνει βεβαίως ε, να είμαστε ανοιχτοί ως προς την έκβαση της συζήτησης. Υπόθηκε ότι με την ενίσχυση των ιδίων πόρων θα απλοποιηθεί η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Βεβαίως, έτσι, υποθέτουμε ότι ένα τμήμα της συζήτησης, δηλαδή το ύψος του προϋπολογισμού, θα παραμεριστεί. Γιατί βεβαίως ένα θα έπρεπε να είναι σαφές ότι αν καθορίζουμε το ύψος του προϋπολογισμού με βάση των ίδιων πόρων, τους ίδιους πόρους, αυτό θα έπρεπε να είναι και το ύψος των δαπανών. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το είδος και το ύψος των δαπανών. Διαφορετικά θα διαπιστώσουμε πάρα πολύ εύκολα πως υπάρχουν διάφορες επιθυμίες, διάφορες ιδέες, μπορεί να είναι καλές, αλλά δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Οπωσδήποτε, εντός του Κοινοβουλίου, θα πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστούμε σε κάποια πράγματα και κάποια άλλα να πούμε «ε, ας τα αφήσουμε κατά μέρος». Δηλαδή βλέπω έναν κίνδυνο εδώ πέρα να πάμε σε έναν αυτοματισμό να ξοδεύουμε συνεχώς περισσότερα λεφτά. Και αν σκεφτούμε αυτά τα οποία μόλις ακούσαμε, όλα έλεγαν ότι όλες οι παρεμβάσει είναι ότι έχουμε κάποιες καλές προτάσεις που πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε και δεν φτάνουν τα λεφτά. Είναι φυσιολογικό νομίζω να μην φτάνουν τα λεφτά για να καλύψουν όλες τις επιθυμίες μας. Πάντα υπάρχουν νέες επιθυμίες. Σας πάρουμε το παράδειγμα της πολιτικής του ασύλου. Γιατί και εκεί πέρα ακούστηκε ότι οι δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν κάποια προσθέμενη αξία και νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ε, πράγματι υπέρ της θέσης ότι για τον τομέα αυτής της πολιτικής χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια της ενός. Αλλά πάντα τονίζω θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική ασύλου που θα λειτουργεί. Πού είναι αυτή, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Οπότε πριν μιλήσουμε για χρηματοδότηση πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε την βάση γι' αυτό. Και εκεί πέρα Νομίζω, αν είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το προσπερνάμε. Επίσης, οι δαπάνες στην γεωργική πολιτική πράγματι είναι μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις δαπάνες κάποιου κράτου μέλου στον τομέα, μέλους στον τομέα της γεωργίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να καταγγείλουμε την αλληλεγγύη καθόλου. με ε, Γερμανός, η Γερμανία είναι καθαρός εισφορέας και θεωρώ πως τα λεφτά τα οποία ξοδεύει η Γερμανία έτσι επενδύονται σωστά για να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αναρωτιέμαι όλα αυτά τα οποία χρηματοδοτούμε μέσω Βρυξελών αν θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται έτσι. Γιατί δημιουργούμε μια περιττή γραφειοκρατία. Γι' αυτό αναρωτιέμαι συχνά τι θα ήταν μια σωστή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε το τι πρέπει να χρηματοδοτούμε και για το τι πρέπει να είναι αρμόδια. Και όταν απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, περνάμε στο αν υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης από τις τωρινές. Θεωρώ πως εάν βιαστούμε και αρχίσουμε τα ζήτω κτλ, θα ε, προσπεράσουμε ένα κομμάτι της συζήτησης και θα πάμε κατευθείαν στους ίδιους πόρους. Αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό για την κριτική ανάλυση που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι πρέπει τελικά να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σταρά. Λόγω έχει κύριο Σταρά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μόντι, κύριε Λαμασούρ και τους υπόλοιπους ε, που συνέταξαν αυτή τη σημαντική έκθεση. Να σας πω ένα μυστικό. Είναι πραγματικά περιζήτητο. Το πήραν από την θηρίδα μου και ζήτησα από τη, βοηθή μου να, από τη βοηθό μου να το κλέψει από έναν άλλο βουλευτή που δεν είναι μέλος της Επιτροπής Οπότε είναι Περιζήτω και αξίζει να το διαβάσουμε. Και ε, καθυστέρησε λίγο, εντάξει. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια θεωρητική έρευνα ως ιδέα, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς έναν απευθείας δεσμό με τους πολίτες. Και ε, βεβαίως πιο σημαντικός, ένας από τους πιο σημαντικούς δεσμούς ε, για τους πολίτες είναι η πληρωμή των φόρων. Γι' αυτό ε, λέω εγώ ότι πρέπει να ενταχθούν σε μια διαδικασία οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, γιατί τώρα πληρώνουν φόρους στα κράτη-μέλη και μετά τα στέλνουν τα κράτη-μέλη κτλ. Έτσι λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα γίνεται αντιληπτή ως ε, ένα κοινό μας ε, έργο, όχι κάτι το οποίο κάνουν κάποιοι στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο ή κάπου άλλο. Γι' αυτό μου άρεσε η στο βερολινο η καπου γι αυτο μου αρεσε η προταση για τον ΦΠΑ που επίσης ε, συζητιέται εδώ και καιρό και ένα ερώτημα θα ήθελα να κάνω. Λάβατε υπόψη μήπως ε, το πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα ενός ε, τέτοιου φόρου γιατί θα υπάρχει βέβαια κριτική ότι θα έχουμε επιπλέον βάρη στους ε, φορολογούμενους και τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για αυτόν τον δεσμό ε, μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να γράφουν οι αποδείξεις Ευρωπαϊκός ΦΠΑ επάνω. Ευχαριστώ κύριε Τάβα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ε, γίνει συμπαθητικός ο φόρος κατανάλωσης για τους συμπολίτε μας. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά πραγματικά θα άξιζε μια σωστή συζήτηση. Ο κύριος Γκάια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την ομάδα εργασίας και, και να συγχαρώ και εσάς κύριε Μόντι. Θαυμάσιο αποτέλεσμα. Περιέχει πολλές προτάσεις και ευχαριστώ και τους τρεις εκπροσώπους μας. Τον συνάδελφο Φερκόφστατ που είναι ακόμη συνάδελφός μας και τον ε, πρώην συνάδελφο Κάλφιν και τον συνάδελφο Λαμασούρ. Νομίζω ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας το αποτέλεσμα αυτό. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το αποτέλεσμα μετά από μια πρώτη ματιά που του Τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε πολιτικά. Αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον χρονικό περιθώριο. Νομίζω ότι δεν ευχαρίστησα τους Βρετανούς ε, συναδέλφους ε, όταν τους είπα ότι βεβαίως ε, κανέναν δεν ωφελεί η αποχωρησή σας, αλλά τουλάχιστον θα διευκολύνει τη διαδικασία απόφαση του προπολογισμού. Πέρυσι είχαμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό, πέρυσι αρχές του χρόνου, ήταν παρόν ο Γερμανός Υπουργό ε, Οικονομίας, ο οποίος είχε πει ότι βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα, αλλά επίσης ε, είπε ε, ότι θα παρέμεναν θεωρητικά τα αποτελέσματά σας, διότι θα τα σταματούσαν οι Βρετανοί άρα δεν θα ήταν ρεαλιστικά. Τώρα που είναι σαφές ότι θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα θα πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί είτε ο κύριος Σόιμπλε και άλλοι υπουργοί οικονομίας θα πούνε ότι ναι βεβαίως πρέπει να το συζητήσουμε ή θα διαπιστώσουμε ότι τελικά κρυβόντουσαν πίσω από τους Βρετανούς μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα. Τώρα θα καταλάβουμε εάν θέλουν να κάνουν κάτι ή όχι. Θαυμάσια έκθεση. Και προσπαθεί να κάνει με σωστό τρόπο τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Να τη βασίσει σε αντικειμενικά στοιχεία. Έτσι, να βγάλουμε τα τοξικά στοιχεία από αυτή τη συζήτηση. έχω ακούσει από υπαλλήλου του δικού μου Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η συζήτηση αυτή γίνεται όπως μας βολεύει. Όταν συζητάμε για ίδιους πόρους μα λένε «Μα τι θέλετε, έχετε ίδιους πόρους, έχετε τους πόρους που σχετίζονται με το ΑΕΠ, έχετε δικαίωμα να αξιοποιήσετε αυτούς τους πόρους, να το αρνούμεθα και κλείνει κάθε περαιτέρω συζήτηση για ίδιου πόρου. Όταν όμω συζητάμε για τι πολιτικέ προοπτικές, και για τον ε, προπολογισμό, τότε λένε μα όχι είναι δικά μας τα λεφτά. Και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν στο δικό μας, το γερμανικό προπολογισμό. Άρα τώρα έχουμε μεγάλες δυνατότητες κάτι να κάνουμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε αυτή η ζήτηση να μην ωφελήσει τελικά τους ε, ευρωλαϊκιστές γιατί αυτή η σύνδεση τους ε, διευκολύνει. Δεν ε, άκουσα κανέναν από αυτούς από το EFDD και το ENF που πάντα επικρίνουν ε, τις ευρωπαϊκές μας ε, προσπάθειες και αυτό με εκπλήσει. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να καταφέρουμε είναι να αποδείξουμε ότι δεν θέλουμε επιπλέον φόρους ε, για τους φορολογούμενους είναι ότι θέλουμε να γίνει ανακατανομή, απλούστευση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προπολογισμού και δεν ανησυχώ όσο ο συνάδελφος διότι από ό,τι κατάλαβα το ανώτατο όριο αυτών που μπορεί να κάνει και χρηματοδοτήσει η Ένωση θα καθορίζεται από κοινού από τα θεσμικά όργανα. Και εάν έχουμε περαιτέρω ίδιους πόρους όπως προτείνεται, τότε φυσικά οι, οι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΠ θα ε, μειωθούν. Είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Οπότε οι εθνικοί προπολογισμοί θα είχαν περισσότερους πόρους. Άρα η τελική σούμα δεν θα είναι ουσιώδης φορολογική επιβάρυνση. Κάτι άλλο. Το ανέφερε και ο Ζωζέ Μανέο. Έχουμε ήδη ένα πίνακα με το κόστος της έλλειψης Ευρώπης, της μη Ευρώπης. Έχουμε κάνει μία απαρίθμηση του τι σημαίνει ο προϋπολισμός της Ένωσης. Ο Αλέν Λαμασούρ μίλησε για τις πρεσβείες. Για παράδειγμα το σύστημα αδειοδότησης φαρμάκων. Άλλο παράδειγμα ένας, ε, μία φαρμακοβιομηχανία, είτε δική μας, είτε ευρωπαϊκή, είτε αμερικανική, είτε ιαπωνική, κάνει μία αίτηση για άδεια, για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά και έτσι αποφεύγει 28 εθνικές αδειοδοτήσεις για ένα φάρμακο. Αν όλα αυτά τα παρουσιάσουμε, αν θυμάμαι σωστά την μελέτη που τα παρουσιάζει, τότε φτάνουμε σε ένα ποσό 100 δις ωφέλους. Είναι απόλυτα σωστό. Πάντα πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά στη συζήτηση. Να τονίζουμε ότι βεβαίως έχει κόστος η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Α, και ότι αυτό που θέλουμε είναι αυτό να γίνεται με διαφανή, με ωφέλιμο, με αποδοτικό τρόπο, με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και πολύ σημαντικές εξοικονομήσεις. Αυτά τα δύο σημεία πρέπει να τα τονίσουμε. Αυτό είναι το κοινό καθήκον όλων όσων θα συνταχθούν με αυτές τις προτάσεις και μόνο έτσι θα έχει αποτελεσματικότητα η έκθεση Μόντι και πρέπει να απευθυνθούμε και στα μέσα, να τους παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Όταν θα λήξει λοιπόν αυτή η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, όπως το λέμε στη Γερμανία, όταν γίνονται όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις δηλαδή για τους ε, προϋπολογισμούς και για τις προοπτικές, όταν όλοι τσακώνονται για το πόσα θα δώσω, πόσα θα κρατήσω, αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση και η έκθεση Μόντι μας το επιτρέπει αυτό, τότε νομίζω ότι αυτό σημαίνει πως και οι δημοσιογράφοι θα έχουν λιγότερη δουλειά να κάνουν και αυτό θα το εκτιμήσουν. Ευχαριστούμε. Αληθεύει αυτό που λέτε. Πρέπει να σταματήσουμε να φρενάρουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να βρούμε και που είναι ο... τα μπραγιάζ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Τούμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα κύριε Μόντι και είμαι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου πολύ ειλικρινά και θα σας ομολογήσω ότι έκανα λάθος. Εγώ δεν πίστεψα. Ήμουν ε, ιδιαίτερα επιφυλακτική πρέπει να πω. Και το αναγνωρίζω ενώπιόν σας. Το αποτέλεσμα είναι πέραν κάθε προσδοκίας και οι προβλέψεις δικές μου διαψεύστηκαν. Συγχαρητήρια λοιπόν και ευχαριστούμε για αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι το έγγραφο που μας προσιάζεται θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε μια πολιτική συζήτηση και ειδικότερα με τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως είπατε. Ε, το είπατε πολύ από εσάς και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό διότι εκεί πιστεύω θα ξεμπλοκάρουν τα πράγματα. Ε, παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι λίγο πιο επιφυλακτική για το κατά πόσο θα ξεμπλοκάρουν τα πράγματα σε επίπεδο συμβουλίου, γιατί όπως ξέρετε για το πολιτισμό στο νομικό πλαίσιο και την αναθεώρησή του, ε, μετά από πολλές συζητήσεις με το Συμβούλιο, όπου θελήσαμε απλά να αναφέρεται στα παραρτήματα το ζήτημα των ιδίων πόρων για το επόμενο, ε, για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και δυστυχώς ε, δεν έγινε δεκτό αυτό. Παρότι λοιπόν ε, ένα κομμάτι έχει συμπεριληφθεί στο ε, έγγραφο και έχει υπογραφεί από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, πιστεύω ότι η ομοφωνία, η όρεξη του Συμβουλίου να ασχοληθεί με τους ίδιους πόρους δεν είναι τόσο μεγάλη, οπότε θα αναγκαστούμε να περάσουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε λοιπόν και για τα κριτηρία που απεριθμίσατε τον κάθε ιδιοπόρο με την ιδέα της ισότητας, της δημοσιονομικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας κτλ. Αρχές που μας βρίσκουν σύμφωνους και που μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτούμε μια εικόνα του κάθε πόρου για να ξέρουμε ποιο τι προτιμάμε σε κάθε πόρο. Αυτό θα χρησιμεύσει ιδιαίτερα στις μελλοντικές συζητήσεις και θα αποτελεί σημαντικό οδηγό. Τώρα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια, διότι το θέμα αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό, πιστεύω για όλα τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Γιατί, διότι μέσω αυτού του ζητήματος θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τρία προβλήματα. Όπως είπατε κύριε Λαμασούρ, ε, το ζήτημα της επικουρικότητας, Και συμφωνώ με κάποια σχόλια, όπως του κ. Κέλμελ, όπου είπαμε ότι όλα αυτά είναι μια χαρά εφόσον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν αρκεί αυτό, ε, Ξέρετε, μιλήσατε για τους συνοριοφύλακες. Δεν πιστεύω ότι τα πρόστα μέσα που διαθέσαμε ε, ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Αν λοιπόν από τη μια πλευρά αυξάνουμε τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταργούμε πράγματα σε εθνικό επίπεδο, δεν δημιουργούμε άριστε συνθήκε. Ωραία λοιπόν, ναι, δημοσιονομική επικορικότητα να ε, τη χρησιμοποιήσουμε ως μέσο για να προχωρήσουμε μπροστά, εφόσον όλα αυτά γίνονται αποτελεσματικά και με επάρκεια. Ε, ο δεύτερος λόγος, ε, όπως είπε η συνάδελφος, είναι το, η ποσότητα θα παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο, γιατί αν παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στα διακυβεύματα, το ξέρουμε πολύ καλά. Και τρίτο σημείο που είναι το πιο σημαντικό, παραδόξως, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο που τα πράγματα έχουν μπλοκάρει, μπαίνουμε σε μία περίεργη λογική, όπου ο κύριος πόρος που κυριαρχεί επί όλων των άλλων, για τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι η εθνική συμμετοχή η οποία αναπόφευκτα οδηγεί σε δημοσιονομική συρρήκνωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για αύξηση. Μιλάμε για τι επίπεδο θα έχουμε, οπότε η κατάσταση οδηγεί σε διέξοδο. Και μετά θα ήθελα κάποιες διευκρινήσει. Όλο λέμε οι ίδιοι πληρώνουν διαρκώ. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Ιβάλλο που ανέφερε αυτό το σημείο, διότι το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι ακριβώς το να μην πληρώνουν πάντα οι ίδιοι. Και όταν αναφέρετε όλα αυτά τα κριτήρια για την ε, δημοσιονομική δικαιοσύνη, ισότητα, όπως την ονομάσουμε, το πρώτο κριτήριο, όταν αναφέρετε όλα αυτά, αυτό είναι ένα μέσο λοιπόν για να, για να βγούμε από το διέξοδο και για να κάνουμε πιο προσφυλές το, το θέμα αυτό. Γιατί ξέρετε, είναι ένα θέμα που δεν είναι προσφυλέ από τη φύση του. Θα κάνουμε τη συζήτηση, αλλά ξέρετε, το ζήτημα είναι το εξής, Το ερώτημα είναι το εξή για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία οι φόροι θα μπορούσαν να γίνουν προσφυλίες στους πολίτες Ναι, υπάρχουν ξέρετε διότι αν δεν έχουμε μαζί τους πολίτες μαζί μας με το πλευρό μας δεν θα περάσουν τα πράγματα δεν πρόκειται να περάσει από το Συμβούλιο Εμέσω μπορεί να περάσουν από το Συμβούλιο, αλλά θα χρειαστεί να περάσουν πρώτα από του πολίτε. Οπότε πρέπει να βρούμε συμπαθεί φόρου. Υπάρχουν τέτοιοι φόροι. Να μην παρατείνω τώρα τη συζήτηση. Οπότε να έχουμε επαναπροσδιορισμό ε, το, όχι μόνο των δαπανών αλλά και των εσόδων. Ε, να δούμε πώς θα αποκτήσουμε νέα έσοδα. Η συζήτηση βέβαια βρίσκεται ακόμα στην αρχή της, οπότε δεν θα παραταθώ. Αλλά μια ερώτηση προς τον κύριο Μόντι και προς τον πρόεδρο τον κύριο Αρτουή. Τι έπεται άμεσα. Διαδικαστικά, ε, τι προοπτικές υπάρχουν, έχουμε μια έκθεση ήδη της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τον κ. Λεβαντόφσκι και τον κ. Ντεπρέ. Έχει ξεκινήσει ο διάλογος με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ενδεχομένως και πέραν των Εθνικών Κοινοβουλίων με τους συμπολίτε μας με το Συμβούλιο και φυσικά στρέφομαι τώρα προς τον ε, αγαπημένο μου συνεισηγητή. Έχουμε και την προετοιμασία του επόμενου δημοσιονομικού, πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, οπότε έχουμε διάφορα εργαλεία στα χέρια μας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, πώς θα... Τα ε, δημιουργηθεί, πώς θα εκπονηθεί όλη αυτή η ατζέντα για το μέλλον. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστούμε, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τους συμπαθείς δίκαιους φόρους, αλλά θα χρειαστεί να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Κύριε Μανκά, έχετε το λόγο, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μόντι, εσείς και τα μέλη της ομάδας σας κάνατε εξαιρετική δουλειά δημιουργήσατε μια θετική ατμόσφαιρα εδώ, κατά το οποίο από μόνο του είναι κάτι το θετικό. Διάσα χθε το βράδυ την έκθεση, έλαβα ένα αντίγραφο και εξαφανίστηκε, ελπίζω να μην ξέρει ο κύριος Τάραντ τι έγινε, όχι αστείευα Λοιπόν, θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες, ε, αλλά χαίρομαι μπορώ να πω ότι συντάσσοντας την έκθεση χρησιμοποιήσατε πληροφορίες από Σλοβάκους επιστήμονες από την Ακαδημία Επιστημών, από το Ινστιτούτο της Βιέννης και χαίρομαι που βρήκατε ένα νέο τρόπο συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ελπίζω τα θεσμικά όργανα να είναι επίσης ικανοποιημένα με αυτόν τον τρόπο για να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια. Αναφέρατε επίσης ε, το ότι δημιουργούνται εμπόδια από τις εθνικές διαδικασίες, ε, π.χ. σε διάφορους τομείς. Ε, ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό. Επίσης, μειώνουμε εμείς τον αριθμό του προσωπικού κατά 1%. Οι Ευρωπαίοι πολίτες το βλέπουν. Αλλά τι γίνεται μετά, για να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση απολύουμε διερμηνείς που τους χρειαζόμαστε και μετά προσλαμβάνουμε εξωτερικούς. Και αυτό παρουσιάζεται ως επίτευξη ενός στόχου. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αν είμαστε πιστευτοί και αξιόπιστοι, πρέπει να είμαστε λογικοί και ειλικρινείς. Είπατε ότι το Συμβούλιο ήταν εναντίον ε, των ίδιων πόρων, ενώ το Κοινοβούλιο τους στήριξε. Μετά παρουσιάστηκε μια γνώμοδότηση που λέει ότι όταν εγκριθούν οι ίδιοι πόροι δεν θα επηρεαστούν οι περιπολογισμοί. Ε, πρόκειται περί λάθους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έτοιμοι γιατί υπάρχει αντίσταση απέναντι σε αυτές τις λύσεις ακόμα και αν είναι σωστές ε, έτσι έχει η ζωή οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι ανάλογο με το δικό σας κύριε Μόντι λοιπόν καλή τύχη εύχομαι και ελπίζω τελικά να επιτύχουμε Ευχαριστώ επειδή έχει περάσει και ώρα να κάνω και εγώ μια ερώτηση ο προϋπολογισμός είναι οι πόροι ε, που αξιοποιούμε για να εφαρμόσουμε μια πολιτική. Άρα το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε, τι πολιτική θέλουμε να εφαρμόσει η Ένωση και τι ε, αρμοδιότητες είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στην Ένωση. Γιατί θα διαπιστώσουν ότι τώρα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν τα κράτη-μέλη δυνατότητα να ασκήσουν ορισμένου τομεί πολιτική και ότι μεταφέροντάς τη στην Ένωση θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε μια γνήσια κυριαρχία αποτελεσματική. Θεωρείτε ότι αν υπήρχαν τέτοιες μεταφορές κυριαρχίας, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική η ευρωπαϊκή κυριαρχία, τα κράτη-μέλη θα έκαναν οικονομίες. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν αντίστοιχα να χρηματοδοτήσουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό με το κόστος της πολιτικής που δεν θα κάνουν διότι ε, είναι σαφές ότι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ασκείται πιο αποτελεσματικά αλλά και με περισσότερες εξοικονομήσεις ε, κάποιος, το, ασκούνται κάποιοι τομείς πολιτική, καλύτε, πολιτικής καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ ενθαρρυντική. Ε, πραγματικά ξεπερνά τις προσδοκίες μου. Και ευχαριστώ και σας ε, και τους βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια και να τονίσω ακόμη μια φορά ότι ήταν ε, συλλογική εργασία. Οφείλω να επανέσω τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο και από τα άλλα θεσμικά όργανα και χαίρομαι που βλέπω εκεί απέναντι τα μέλη της γραμματείας που έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και γεγονός είναι ότι πράγματι περιλάβαμε διάφορα επιστημονικά ιδρύματα και think tank γιατί είναι πολιτική έκθεση αλλά γνωρίζουμε εκ ότι θα την πάρουν σοβαρά μόνο εάν έχει πολύ στιβαρή αναλυτική και τεχνική βάση. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου μια εξομολόγηση προς την κυρία Τόμα. Πρέπει να ομολογήσω και προς την Επιτροπή σας γενικότερα ότι ένα μυστικό κίνητρο του έργου μου στην ομάδα αυτή ήταν να πίσω την κυρία Τομά και να την ε, καταφέρω να ξεπεράσει την έλλειψη εμπιστοσύνης ε, στο αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Ελπίζω λοιπόν αυτή η αμοιβαία αναγνώριση ε, η αρχή αυτή της ε, Ένωσής μας να αποτελεί καλόν ιονό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σύντομα σε κάποια ζητήματα που αναφέρθηκαν και βεβαίω με ευχαριστώ ε, και ο Αλέν και άλλοι συνάδελφοι να συμπληρώσουν τις παρατηρήσεις μου ένα ενδιαφέρον σημείο και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές, τους μόνους εισηγητές και τους συντονιστές. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής. Ίσως λόγω των δύο αυτών στοιχείων των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών και του Brexit ε, μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ίσως και νωρίτερα από όσο περιμέναμε για να αντισταθμίσουμε ακριβώς αυτές τις ελλείψεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πιθανώς έχει... είναι λογικό. Ταυτόχρονα, επειδή ε, είναι ήδη μπορεί πόροι, είναι κάτι το νέο, ίσως απαιτηθεί περισσότερος και όχι λιγότερος χρόνος για να γίνει τη προετοιμασία και εφαρμογή. Ίσως θα μπορούσαμε. Κάποιοι νέοι πόροι που θα λαμβάνουν την μορφή προσθήκης σε υφιστάμενες μορφές φορολογίας στα κράτη-μέλη να συνδυάζουν την άμεση εφαρμογή καθώς δεν θα χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μια ιδέα έτσι. Και... Συμφωνώ ότι θα μπορούσε βεβαίω να είναι μια γενική αρχή ότι οι πόροι αυτοί που προκύπτουν από κοινοτικές αρμοδιότητες ε, θα μπορούσαν επί της αρχής να είναι αφιερωμένοι στον κοινοτικό προπολογισμό. Είμαι σίγουρος ότι ε, τα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρατε ε, θα μπορούσε να έχει το να βασιστούμε στον ΦΠΑ νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα απαντήσουν οι συνάδελφοι που έχουν μεγαλύτερη πείρα στον ΦΠΑ κάποιος είπε σε μια παρέμβαση παρά το ότι εξέφρασε θετικές απόψεις για την έκθεσή μας και τον ευχαριστώ είπε ότι καθυστέρησε η έκθεση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, κοιτάξτε, χρειάστηκε χρόνος για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, αλλά νομίζω πως ήταν ε, σοφή απόφαση των τριών θεσμικών οργάνων όταν προετοίμασαν την εντολή για την έκθεσή μας το 2014, αρχές του 2014 και έθεσαν ως προθεσμία το τέλος του 2016 αρκετά άνετο χρονοδιάγραμμα και νομίζαμε ότι βεβαίω. θα ήταν επικίνδυνο και κάπως έτσι μια ένδειξη και αλαζονίας από μέρους μας ε, ολοκληρώσουμε την έκθεση πριν από την προθεσμία. Και τελικά αποδείχθηκε ότι συνέβησαν τόσα πράγματα στο τελευταίο έτος της προθεσμίας, έτσι ώστε αν είχαμε ολοκληρώσει την έκθεση στα μέσα ή στο τέλος του 2015, που θα ήταν τεχνικά εφικτό, δεν θα ήμασταν σε θέση να εκφράσουμε απόψη για τις επιπτώσεις του Brexit για την σχέση μεταξύ των πτυχών του προϋπολογισμού και της ε, νέων αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως π.χ. μετανάστευση κτλ. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τα τρία θεσμικά όργανα. Όχι τόσο επειδή μας έδωσαν μεγάλο χρονικό περιθώριο, αλλά επειδή προέβλεψαν ένα χρονικό διάστημα το οποίο είχε τόσα πολλά ευχάριστα και δυσάριστα γεγονότα και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζουν το θέμα μας. Γρήγορα κάτι για την ερώτηση του ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί. Αυτό νομίζω θα το απαντήσει ο πρόεδρος ο κύριος Αρτουή, αλλά προσωπικά και οι συνάδελφοι επίσης νομίζω θεωρούμε ότι θα πρέπει τώρα να υπάρξει κάποιο είδους ε, ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, προς την κοινή γνώμη, προς τα θεσμικά όργανα για την έκθεση αυτή, να γίνει μια δημόσια συζήτηση και νομίζω μπορείτε να βασίζεστε πάνω μας αν θεωρείτε κάτι τέτοιο αναγκαίο. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω, οπωσδήποτε, όπως είπε κάποιος από εσάς, ε, υπάρχουν ακόμα εκλογές σε πολλά κράτη-μέλη που ίσως αποτελέσουν εμπόδια για την σοβαρή συζήτηση αυτών των θεμάτων, αλλά αυτό είναι αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ σε μια δημόσια ενημερωτική συζήτηση. Εγώ θα ζητούσα από προέδρους κυβερνήσεων και ε, υπουργούς οικονομικών το εκλογικό τοπίο, για να μην μιλήσω για τα δημοψηφίσματα, έχει γίνει πολύ προβληματικό στην Ένωση και είναι εκρηκτικό το να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωτερική πολιτική συζήτηση. Και πολλά από τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση έχουν το πρόβλημα του πώς να αντιμετωπίσουν το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με τα ευρωσκεπτικιστικά, εθνικιστικά και κόμματα. Ε, ε, μ' αρέσει η λέξη λαϊκιστικά. Ίσως αυτοί οι αρχηγοί κυβερνήσεων θα μπορούσαν να σκεφτούν το εξής και οι Υπουργοί Οικονομικών. Προσπαθούμε προσελκύσουμε ψυχοφόρους από τους ε, ευρωσκεπτικιστές, ε, τους ε, εθνικιστές, μέσω της οικονομικής γενεοδορίας. Δηλαδή προσπαθούμε όπου είναι δυνατόν να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη κτλ. για να κερδίσουμε τουλάχιστον κάποιους ε, πόντους εκεί στην αξιολόγηση των ψηφοφόρων. Αλλά θα έπρεπε ίσως να σκεφτούν ότι ο λόγος για τον οποίο σε πολλές χώρες, πολλές εκλογές ε, και πολλοί ψήφοι πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα, ε, ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση με τις αυστηρά οικονομικές στοιχές, ε, το επίπεδο φορολογίας ή της αγοραστικής δύναμης, αλλά πλέον έχουν περισσότερη σχέση με πιο θεμελιώδεις ανησυχίες και φόβους για την μετανάστευση, τους πρόσφυγες, την τρομοκρατία, την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και θα έλεγα στους υπουργούς και πρωθυπουργούς πως αυτά είναι δημόσια αγαθά τα οποία δεν αγοράζονται στο σούπερ μάρκετ με υψηλότερη αγοραστική δύναμη και εσείς πάντα λέτε ότι εσείς τα κράτη-μέλη δεν μπορείτε πια να παρέχετε αυτά τα δημοσία αγαθά τα οποία θα βελτιώσουν την πραγματική κατάσταση των πολιτών γιατί θα αισθανθούν πιο ασφαλείς σε μια έτσι, έφτακτη συμφωνία, ε, κοινωνία αλλά ίσως είναι προς ε, το συμφέρον σας και το εκλογικό σας συμφέρον να σκεφτείτε πώς θα πρέπει να επιμείνετε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ίσως η μόνη οντότητα που μπορεί τελικά να παρέχει αυτά τα αγαθά που θέλουν ε, απεγνωσμένα οι πολίτες. Αν λοιπόν θεωρείτε πως κάποιες τέτοιες αρμοδιότητες ανήκουν αναπόφευκτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο Ίσως ε, μπορείτε να κάνετε και το τελευταίο βήμα και να πείτε ότι αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και αξιόπιστοι, ε, νέες ε, αρμοδιότητες σημαίνουν και νέους ιδίους πόρους. Οπότε θεωρώ ότι έτσι οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός προπολογισμού ο οποίος θα βλέπει και το μέλλον δεν θα πρέπει να είναι τόσο δειλή ε, θα πρέπει να έχουν μια νοοτροπία που θα κοιτάει προς το μέλλον και ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάσουν την έκθεση προσεκτικά πράγματος χάρη η σημερινή Handelsblatt στο διαδίκτυο γράφει ένα σχόλιο κάποιο τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σπαν, τον ε, Υφυπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, που ρωτήθηκε για την αντίδραση της ε, Γερμανίας στην έκθεσή μας και είπε γρήγορα ότι είναι τελείως ε, άχρηστη. Το θέμα δεν είναι περισσότερα λεφτά για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά η καλύτερη χρήση των πόρων. Θεωρώ ότι μια ακριβής ανάγνωση της ε, έκθεσής μας θα καθησυχάσει τις ε, ανησυχίες ε, του κυρίου αυτού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο στην συνέντευξη τύπου που ε, Αλάν Λαμασούρ. Euh, le président Monti a, a répondu l'essentiel des questions. Deux ou trois points. D'abord, Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Ε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα ε, συγχαρητήρια και ας μην ξεχνάμε την Αλμοτανιό που ε, ανέλαβε τη σύνταξη του εγγράφου, έγραψε το έγγραφο και βρίσκεται εκεί πίσω πίσω κάθεται μια εξαιρετική συνεργάτης του Μάριο Μόντι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ηγήθηκε της ομάδας ε, και βοήθησε την ε, ε, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Ο Μαρίο Μόντι απάντησε και συμφωνώ στο πολύ έξυπνη παρατήρηση δεν μας εκπλήσει η ευφυΐα βέβαια του Ζεράρ Ντεπρέ που είπε αφού αποφασίσουμε ευρωπαϊκή πολιτική που να συνεπάγεται δημιουργία δημοσίων δαπανών θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκό στόχο Και εδώ χάσαμε μια καταπληκτική ευκαιρία. Και εγώ είμαι υπεύθυνο γι' αυτό. Ε, Ω χριστιανοδημοκράτη, μάλλον θα περάσω χρόνια και χρόνια στο καθαρτήριο γιατί. Ε, μάλλον θα πάρετε. Μάλλον είναι πλεονέκτημα αυτό. Ε, χάσαμε την ευκαιρία του ETS, δηλαδή τον πληστηριασμό των ε, δικαιωμάτων να ρηπαίνει κανείς, έτσι το λέμε στην καθομιλουμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στι πρώτε αξιολογήσει είχε κάνει λάθο διότι ήταν κακοσχεδιασμένο το αρχικό σύστημα, αλλά είχε προβλέψει 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίω έσοδα από αυτά και ξαφνικά έχουμε μια ευρωπαϊκή ε, νομική βάση για μια αγορά ε, δικαιωμάτων για ρήπανση ευρωπαϊκών και στο επίπεδο του Συμβουλίου θεωρείται ότι αυτό αυτόματα θα τροφοδοτούσε τους εθνικούς ε, προπολογισμού και κανείς δεν αντέδρασε. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να ε, δώσατε ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Η που είναι αυτό η ένωση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μελετά μια ε, ε, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σενάριο, θεωρώ εγώ, που συνίσταται στο εξή. Λέει ότι όλα τα προβλήματα που θα εμφανιστούν, κυρίω τα προβλήματα των νέων τεχνολογιών, ε, που θέτουν νομικά, νομικά θέματα όπως η βιολογία, θα πρέπει να εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το μέλλον και να μην δηλητηριάζουμε το μέλλον με 28 διαφορετικά συστήματα. Για παράδειγμα, ε, η ψηφιακή τεχνολογία. Δεν μπορούμε να έχουμε 28 εθνικές νομοθεσίες για την προστασία των ψηφιακών δεδομένων. Και με προλάβετε το είπατε, οι Βρετανοί φίλοι κάποια στιγμή ανέφεραν τη δυνατότητα να επιβληθεί φόρο στο Google. Ε, δεν έγινε αυτό, αλλά δεδομένων των συγκεκριμένων ε, ε, πολύ ευαίσθητων προβλημάτων του ψηφιακού κόσμου, δεν μπορούμε να έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα. Και μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω για αυτό το ε, θέμα όσον αφορά την αναρμόνιση της φορολογικής βάσης για τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων. όπως έχουμε κάνει εδώ και 30 χρόνια για την ε, βάση για το ΦΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πολυάριθμες προτάσεις του Κοινοβουλίου και μετά από το σκάνδαλο LuxLeaks παρουσίασε ένα σχέδιο εναρμόνισης που που ονομάστηκε με το αγγλικό αγρόνιμο CCTB με το γαλλικό αξίς ε, και στις προτάσεις που κάναμε δύο εισηγητές ε, αναφέρεται αυτή που λέει το εξής αφού εναρμονίσουμε τις βάσεις ορισμένων κρατών για ορισμένους φόρους, όπως συμβαίνει ήδη με το ΦΠΑ, όπου προτείνουμε να προσθεθεί ένα ή δύο ε, ποσοστία σημεία στο ΦΠΑ για να τροφοδοτηθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, ε, ε θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με τα κερδί των επιχειρήσεων, να προσθέσουμε ένα ή δύο ε, ποσοστία σημεία μια ίδιο ποσοστία μονάδε μονάδες ε, και εκεί. Φυσικά συμφωνώ με την παρατήρηση της ΕΔΕΡ 1% δεν είναι αρκετό. Απ' τη μια ισχυριζόμαστε ότι έχουμε ε, παγκόσμιε πολιτικές και τις χρηματοδοτούμε τόσο λίγο. Το νέο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας βοηθήσει να πείσουμε από πολιτική άποψη είναι ο πολλαπλησιασμός των ε, δευτερευόντων ε, προϋπολογισμών. Ας δούμε τη συμφωνία με την Τουρκία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού κύματος από τη Συρία. Ε, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα κοινοτικά και δημιουργήσαμε ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται ουσιαστικά από τα ΕΠ, από τις συμβολές συμμετοχές ΑΕΠ των κρατών μελών. Και εκεί έχουμε τον πίνακα που δείξαμε και εκεί έχουμε μία βάση για να μπορέσουμε να πούμε, να σοβαρευτούμε λίγο. Ουσιαστικά οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ μα κοστίζουν πολύ περισσότερο από το 1%. Εάν βάλουμε και όλου παράπλευρου προπολογισμού, χρηματοδοτούνται με τρόπο απόλυτα ασαφή, χωρί κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει, ε, αλλά τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, με τη συμφωνία για την Τουρκία, α πούμε, είπε ο Υπουργό Οικονομικών Γαλλία. Ε, Γαλλίας, ε, εξήγησε στην, ε, ε, στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ότι δεν έχετε παρά να ψηφίσετε ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε πρέπει να επιμείνουμε στο παράδοξο, στο ότι υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι δημιουργούμε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει απόλυτα με ανεπαρκή χρηματοδότηση και που κανείς δεν ελέγχει. Ό,τι χειρότερο δηλαδή να μην επανέλθω στο ΦΠΑ που ανέφερε ο συνάδελφος που δεν είναι πια εδώ ε, αλλά έκανε μια πολύ ε, εύστοχη παρατήρηση. Ευχαριστώ. Υπήρξε πριν από μερικού μήνε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη που υπερεύει τι προσδοκίε όσο με αφορά. Γιατί έχω συμμετάσχει σε πολλέ συνδιασκέψει με συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων που πολύ συχνά δεν είναι καθόλου διατεθειμένα να συζητήσουν αλλαγέ στην νομοθεσία όσον αφορά τη φορολογία. Αυτή τη φορά όμω ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τι διαπιστώσαμε σε αυτή τη διάσκεψη, τουλάχιστον όσοι πήραν το λόγο. Ε, πολλοί σοσιαλιστέ, πολύ καλό αυτό, δεν ξέρω τώρα τι θα έλεγαν όσοι δεν πήραν το λόγο, είπαν λοιπόν ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι επιστροφέ, να απλωστευτούν τα έσοδα ότι το ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να διατηρηθεί αλλά ε, δηλαδή ότι ο ίδιος πόρος ΑΕΠ πρέπει να διατηρηθεί αλλά το ποσοστό να αυξηθεί. Αυτά λέμε και εμείς στην έκθεσή μας και προτείνουμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο για το πώς μπορεί να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να εμπλακούν και τα εθνικά κοινοβούλια που είναι αρμόδια για τις αλλαγές στη φορολογία. Μπορούμε να συζητούμε ό,τι θέλουμε εμείς για τα φορολογικά, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια αποφασίζουν για τη φορολογία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι στο πλευρό μας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από απλές ε, ε, συνδιασκέψεις κάθε τόσο. Πρέπει να έχουμε στο πλευρό μας και τα εθνικά και τα τοπικά κοινοβούλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και όπως θα λέει και η κυρία Τωμά δεν ήξεραν ότι είναι αδύνατο και το έκαναν. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος μιας φάσης. Όλοι έχουμε συνέστηση ότι η Ευρώπη κινδυνεύει. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι το μέσο με το οποίο θα ενημερώνουμε και θα διδάσκουμε τους πολίτες για την Ευρώπη. Περνάτε τώρα σε άλλους τη σκητάλη και τώρα λοιπόν η σκητάλη είναι στα χέρια του, των τριών θεσμικών οργάνων. Και για το Κοινοβούλιο είμαι πεπισμένο και ο εισηγητή Γιάννου Λεβαντόφσκι και Ζεράρ Ντεπρέ θα εργαστούν επ' αυτού. Είμαι πεπισμένο ότι αμέσω θα ασχοληθούμε με την έκθεσή σα στα πλαίσια τη ε, συζήτηση για το επόμενο πολιετέ πλαίσιο. Διότι τα διακυβεύματα είναι πολύ σοβαρά η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλήσει με τους Ευρωπαίους και ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα αδιαφανής. Το καταλαβαίνουν μόνο οι κυβερνήσεις και όχι οι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν και οι πολίτες. Πρέπει να μπορέσουμε να αποδείξουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι υποχρέωσή μας. Να αποδείξουμε επίσης ότι υπάρχει και κοινοβουλευτική προστιθέμενη αξία ότι εδώ δεν κάνουμε σαν να είμαστε κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στις ε, προηγούμενες διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Η επόμενη θα γίνει τον προσεχή Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουάριου. Είναι λοιπόν σημαντικό ήδη από τον επόμενο μήνα στην διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη να συζητήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια την έκθεσή σας. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Μάριο, σε περιμένουν οι δημοσιογράφοι εδώ στους ε, διαδρόμους. Άρα δεν έχει τελειώσει εντελώ η εργασία μας. Θα πρέπει να συνεχίσετε, να τη συνοδεύετε, να μας ενθαρρύνετε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάθε βούληση, κάθε ε, διάθεση και νομίζω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί αποδεικνύουν ότι έχουμε κάθε καλή διάθεση. Και το γεγονό ότι μα λείπουν οι πόροι είναι ε, ακριβώ και ένα κίνητρο για να επιδείξουμε ευφυα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρίασή μα θα γίνει στι 25 και 26 Ιανουαρίου στις 11.45 θα ε, αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Μέχρι τις 12.30.